Dear colleagues, we can start today. Welcome to everybody. If you can... Καλώς ορίσατε όλοι. Καθίστε παρακαλώ. Also, uh, continue in Italian. First... Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. First of all, we have to adopt the agenda. Καταρχήν την ημερήσια διάταξη. Σε siete d'accordo. Συμφωνείτε Ας περάσουμε στην έγκριση της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο σημείο 2. Σήμερα η μέρα μας είναι ιδιαίτερα φορτωμένη, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ελπίζω να έχουμε προσέλευση και το απόγευμα για την ακρόση, για τα εκπαιδευτικά, συστήματα και την απασχόληση των νέων. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν είχαμε αθρώα προσέλευση ε, και το απόγευμα. Δεύτερο σημείο έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων 19-20 Ιανουαρίου, 27 Ιανουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Τρίτο σημείο, μερικές ανακοινώσεις. Σήμερα θα έχουμε διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, δανέζικα, ολλανδικά, ε, ελληνικά, ισπανικά, εστονικά, λιθουανικά, τσεχικά, πολωνέζικα, σλοβένικα, βουλγάρικα και ρουμάνικα. Θα ήθελα επίσης ε, να σας ενημερώσω ότι τη η συνεδρίαση και μία Άλλη πληροφορία θα ήθελα να σας δώσω. Πλησιάζουμε την 8η Μαρτίου. Στις 5 Μαρτίου από τις 9 ως τις 12 έχει ληφθεί μια πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και όπως γνωρίζετε έχει γίνει μια διακοινοβουλευτική συνάντηση με τη συμμετοχή μελών εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια στο χώρο της εκπαίδευσης και το πώς θα μπορούσε να προωθηθεί η συμμετοχή τους. Δεν με παρούσα στην οριζόντια, είμαι παρούσα στην ε, επιτροπή που δημιουργήθηκε. Έχουν προβλεφθεί τρία πάνε. Το πρώτο στη σημασία της εξάλληψης των διακρίσεων μεταξύ των φίλων στον τομέα της εκπαίδευσης. Δεύτερον, πρόκληση για ίση πρόσβαση. Και τρίτον, ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις πτυχές οι οποίες εστιάζονται στο θέμα της εκπαίδευσης και των επιτόσεων που έχει τις γυναίκες. Θα έχω τη χαρά να συμπροεδρεύσω σε αυτή τη συνάντηση από κοινού με την Καρσία Πέρες που είναι πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών. Και βεβαίω θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή αν όλα τα μέλη, άντρες και γυναίκες της Επιτροπής θα μπορούσαν να παραστούν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι στις 28 Ιανουαρίου στην συνδιάσκεψη στην Ολομέλεια είχαμε μια πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας που θα συζητήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής. Όπως θυμάστε, Εστάλει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ως αρμόδια επιτροπή και σε άλλες ε, επιτροπές όπως η Επιτροπή Πολιτισμού για γνωμοδότηση. Στην πραγματικότητα, μια άλλη οργάνωση υπήρξε μια άλλη πρώτα, μια άλλη ε, πρόταση στην διάσκεψη των Προέδρων. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα σε λίγο όταν θα μιλήσουμε για την έκθεση που θα συντάξει ο, ο κ. και εκεί ο ρόλος μας θα είναι πιο σημαντικό. Η γραμματεία ενημέρωσε τις ομάδες και διορίστηκε ο εισηγητής. Η ομάδα του ΕΛΚ είχε μία σειρά από σημεία με βάση το δικό του αίτημα και διορίστηκε, ορίστηκε εισηγητής με γραπτή διαδικασία ο κύριος Δρογεύσκη ο οποίο ειδικό άλλο θα κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Θα επανέλθουμε σε κάθε περίπτωση σε αυτό το σημείο σήμερα. Η μία άλλη πληροφορία. Οι συντονιστέ θα συναντηθούν στο τέλο τη σημερινή συνάντηση τη Επιτροπή για λόγους ε, χρονοδιαγράμματος, είναι πέμπτη σήμερα, οι συστάσεις ε, θα διανεμηθούν σε γραπτή μορφή και συνεπώς δεν θα ανακοινωθούν στην αρχή της ακρόασης. Εάν δεν διατυπωθούν σχόλια μέχρι αύριο το μεσημέρι, θα θεωρηθεί ε, εγκριθήσα η έκθεση των συντονιστών. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα να σας ενημερώσω με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, να περάσουμε στο σημείο 4. Στην έκθεση, με την έκθεση πρωτοβουλία του συναδέλφου Μισελ Ρεϊμόν, επιδίωξε ανανεωμένη συνένεση όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοτική ιδιοκτησία στην εσωτερική αγορά. Είδατε ότι έχουμε ένα πολύ πεπαρημένο χρονοδιάγραμμα, θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια προσπάθεια να περιορίσουμε τις παρεμβάσεις μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι παρεμβάσεις σε λίγα λεπτά και ε, να είναι και κάπως ορθολογικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας. Μετά έχουμε την ψηφοφορία επί αυτής της γνωμοδότησης. Ξέρετε ότι είναι μια γνωμοδότηση για την οποία υπευλήθησαν πολλές τροπολογίες. Η Επιτροπή Γιουρίνη είναι υπεύθυνη για αυτό το ντοσχέ και επιβλήθησαν 49 τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί πράγμα θέλετε να μιλήσετε αγαπητέ συνάδελφε. Α, ο συνάδελφος Θέσος. Θέλετε να πείτε κάτι για τις ε, εργασίες μας. Ο κύριος Γκλέζος. Παρακαλώ. Μικρόφωνο κύριε Γκλέζο. Μόνο ένα λεπτό σας παρακαλώ πριν από την σε διάταξη. Ε, κλείνουν ακριβώς ένας μήνας από τότε που ο ελληνικός λαός εψήφισε για να ανακτήσει την εθνική του ανεξαρτησία και για να βγάλει τη θηλιά που έχουν βάλει στο λαιμό του οι δανειστές. Και το θέμα είναι σημαντικό επειδή είμαστε Επιτροπή Πολιτισμού και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά πολιτισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η δημοκρατία την οποία όλοι προσκυνούμε σήμερα. Θέλω να ειδοποιήσω όλους ότι όλοι όσοι προσπαθούν να μην πετύχουν οι στόχοι και να αναιρέσει ο λαός την ψήφο του θα αποτύχουν. Καλό και ζητώ από όλους τους συναδέλφους υπεύθυνου στον πολιτισμό εάν θέλουν να διατηρηθεί ο πολιτισμός πρώτο και κυριαρχικό σημείο είναι να σεβόμαστε τη θέληση του λαού. Τίποτα άλλο. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ για την έκκληση που κάνετε. Ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα στην χώρα σας. Θα θέλαμε να, να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάθε ελεύθερη φωνή έχει τη δική της βαρύτητα και θα εισακουστεί. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα ήθελα να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Μικέλ Ρέιμον. Θα ήθελα να μου πείτε αν ο εισηγητής θέλει να πει κάτι πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία. No. Όχι. Παρακαλώ. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να πάρω την καρτέλα μου. Succede.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 Σκουζάτε. Ζητώ συγγνώμη. Έχω τόσα πράγματα στο μυαλό μου που ξέχασα την ε, καρτέλα μου. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Παράγραφος 1. Τροπολογία υπαριθμών 1. Μισό λεπτό, να αναφερθώ σε ένα σημείο. Στην παράγραφο 1, τροπολογία 3, η οποία έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία 1, άλλαξε ε, η άποψη του εισηγητή. Ο εισηγητή είναι υπέρ, να σα το πω αυτή εξ αρχή. για να δείτε τι θα κάνετε. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1, παράγραφο 1. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 1, καινούρια. Τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 η οποία τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία. 1. ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 4. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ, ψήφι Συγγνώμη, συγγνώμη. 6. Α, τροπολογία έξι. με συγχωρείτε. Τροπολογία 6, παράγραφος ένα. Είναι ξεχωριστή η ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ, ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ψήφι υπέρ, ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 7, όπως έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 8, παράγραφος 1 σε καινούρια, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο, την καινούργια παράγραφο παράγραφο τροπολογία 9, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 ή νέα, τροπολογία 10, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1F καινούργια. τροπολογία υπαριθμών 11. Να ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 11. Ζήτω. Τροπολογία 11. Τροπολογία. Α, 10. 10. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 10. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Α, το ΕΛΚΑ έχει ένα επιπλέον άτομο. Α, να αφαιρεθούν δύο καρτέλες. Ωραία, ξεκινάει η ψηφοφορία με το σωστό αριθμό μελών. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 18 ψήφους κατά 7 δύο εποχές. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 11. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Για να κάνουμε και έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία υπαριθμών 11. Ίσως έκανα λάθος, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. για να ψηφίσουμε και πάλι, ψηφίζουμε και πάλι την τροπολογία υπαριθμών 11. Πέραση ψηφοφορίας. Ψήφι υπέρ. Τροπολογία 12. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 13 την οποία έχει τροποποιήσει η προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Ψήφι υπέρ, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 14 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 ψήφι υπέρ, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμό 18, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, Νομίζω, νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ποιος εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 22. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 23. Α, μισό λεπτό. 26, περνάμε στην 26. Αν ε, ε, ψήφι υπέρ 26, ψήφι κατά της 26, αποχές εγκρίνεται, 27 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, 28 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, 29 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, Περνάμε στην τροπολογία 30. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 35 η οποία έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία υπαριθμών 4. Ψήφι υπέρ ψήφι κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίθηκε. εγκρίθηκε. Τροπολογία υπαριθμών 36, όπως έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία 5, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37. που τροποποιεί την έξι ψηφί. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 38 πως τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία υπαριθμών 7 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 πως έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία 8 ψήφι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 40 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 41 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, περνάμε στην 43 του κυρίου Γραμματικάκη, Συγγνώ, συγγνώμη, συγγνώμη, ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος, ψηφίζουμε το πρώτο μέρος, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο μέρος, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 του κυρίου Γραμματικάκη, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 πάντοτε του κυρίου Γραμματικάκη, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 46 Μαρλέν Μίτσι, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται 46 Αδεινόλφη ψηφί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μπα. Να κάνουμε μια επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί σηκώστε το χέρι σας Ξεκινάει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 20 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται 49 ε, νέα παράγραφος 5α Μαρκ Ζουλό σελίδα στο κείμενό μου. 48, 48 βεβαίως το ξεχάσαμε αντινόλφη, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται, 49. Παράγραφος 5, η νέα, Μαρκ Ζουλό. Δεν το έχουμε εμείς εδώ όμως. Τώρα είμαστε στο 49. Μάρκ Ζουλό. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως ζητήθηκε για, την, για όλη την έκθεση. Ξεκινάει η ψηφοφορία για όλη την έκθεση. Dichiaro chiusa la votazione. Un attimo, solo votato 22. Sì. Sì. No, dobbiamo rifarlo ancora? Θα πρέπει να ψηφίσουμε και πάλι. Μόνο 22 μέλη εδώ. Υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα. Allora, we repeat the... Ωραία, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Παρακαλώ. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 9 κατά, 2 αποχές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Ρέιμον και συνεχίζουμε στο, με το επόμενο σημείο. Bene, ora abbiamo l'informativa sul παρουσίαση από τον κύριο Σντρογεύσκη της γνωμοδότησης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το λεγόμενο ΕΦΣΙ. Α, κύριε Ρε... Ρέιμον, ζητήσατε το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εδώ βεβαίως συνεργαστήκαμε τους τέσσερις και όλους ηγητές. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Βεβαίως δεν ήταν παρόντες εδώ στην πρώτη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Ευχαριστώ παρόλα αυτά. Καθότι θεωρώ πραγματικά ότι ήταν πολύ σημαντική και η συνεισφορά τους. Κοιτάξτε, δικαίωμά του είναι. Νομίζω ότι έκανε τη δουλειά του και νομίζω ότι και οι συνάδελφοι έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη δουλειά. Τέλο πάντων, είναι δικαίωμά του και ελπίζω στο μέλλον τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Τώρα λοιπόν, όπως σας είπα, ε, περνάμε στην έκθεση Σντρογεύσκη ε, σχετικά με το πρόγραμμα ΕΦΣΥ. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, όπως σας είπα, που έλαβε χώρα στις 10 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε η δική μας Επιτροπή να συνδεθεί με τον κανονισμό 53 συν. Ε, αυτή είναι μια πρακτική που όπως γνωρίζετε ε, θεωρεί αυτή η πρακτική ότι εμείς είμαστε συναρμόδιοι και με άλλες επιτροπές, ε, την ΕΜΠΛΕ, την ΙΜΚΟ, τη ΡΕΤΖΙ, την ΚΟΝΤ μεταξύ άλλων. Άρα δηλαδή οι αρμόδιες επιτροπές για αυτό το σημαντικό νέο ταμείο για τον κανονισμό το σχετικό είναι η ΕΚΟΝ και η budget, budget που είναι με βάση το άρθρο 55, η ΤΡΑ και ΤΡΑΝ με βάση το άρθρο 54 είναι επίση συναρμόδιες. Αν θέλετε δηλαδή συμμετέχουν όλες οι επιτροπές σε διάφορα επίπεδα γιατί η Ήτρα και η ΤΡΑΝ είναι οι επιτροπές εκείνες που έχουν σχέση με εκείνο το κομμάτι του προπολογισμού το οποίο προβλέπει ε, χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις μέσω του προγράμματος Υπότιτλοι AUTHORWAVE Horizon και Connecting Europe. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει πολλή χρόνο. Πρέπει να επιταχύνουμε σήμερα το σχέδιο γνωμοδότηση το έχουμε μόνο στα αγγλικά, αλλά τι τροπολογίε μπορείτε να τι καταθέσετε σε όλε τι ε, γλώσσε. Και ε, οι ε, μεταφράσει μόλι είναι έτοιμε θα σα τι δώσουμε. Τώρα, η ψηφορία στην ECON και στην Budget προβλέπεται στι 20 Απριλίου, εμεί 24 Μαρτίου και η διορία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 11 Μαρτίου μέχρι στις 6 ε, ώρα το απόγευμα. Ε, συνάδελφος Σντρογεύσκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής και επίσης ε, ευχαριστώντας και την πρώην πρόεδρο της Επιτροπής μας, την κυρία Ντόρις Πακ, ε, για την υποστήριξη που προσέφερε στα βραβεία Λουξ και γενικότερα για την υποστήριξή της στον τομέα των ε, κινηματογραφικών ταινιών. Τότε θα θυμάστε επελέγει και η ταινία Ίντα που πήρε και Όσκαρ για τις ξενόγλωσσες ταινίες. Άρα δηλαδή είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που έχει γίνει σχετικά με τα βραβεία Lux. Όσον αφορά τώρα αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που σας ε, κατατέθηκε, πρόκειται αυτό που έτσι πολύ σύντομα λέμε το Ταμείο Juncker, επενδύσεις Juncker. Στόχος είναι λοιπόν οι επενδύσεις, ε, οι στόχοι και η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πώς ε, θα γίνει αυτό, πώς θα ε, επιμερίζονται οι πόροι από αυτό το Ταμείο. Η δική μας Επιτροπή συνδέεται μόνο με τους στόχους του Ταμείου και θα ήθελα να κάνω τα εξή σχόλια. Πρώτα απ' όλα, όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει μία πρωτοβουλία και βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να προαχτεί ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας στρατηγικής. Και αυτή η στρατηγική ε, περιλαμβάνει ε, πόρους ε, ιδεών ε, για να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την χρηματοψηφική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για αυτό το πρόγραμμα που περιλαμβάνει και έναν ε, κανονισμό που θα διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή λέει ότι θα εκταμιευτούν κοινοτικοί πόροι για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις. 16 εκατομμύρια ευρώ θα ε, δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτή με τη σειρά της ε, θα διαθέσει και αυτή άλλα 5 δις ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μιλάει για 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και να αυξήσει τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς με την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε λοιπόν να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και εγώ ε, σε αυτό θέλω να συγκεντρωθώ, στην εκπαίδευση. Βεβαίως δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήρθε σε επαφή με τον πολιτιστικό τομέα και με τον τομέα των δημιουργών γιατί και εκεί υπάρχει δυναμικό ανάπτυξης αυτός ο τομέας είναι άρρηκτα συνδεμένος με διάφορους τομείς ε, της οικονομίας και προσελκύει επενδύσεις. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο πολιτιστικός τομέας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ε, στους τομείς ε, που στοχεύουν στην ανάπτυξη. Εν πάση περιπτώσει το λιγότερο μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να αποκλείεται ο πολιτισμός. Ε, θεωρούμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στην επιτυχία αυτού του προγράμματος. Ε, η χρηματοδότηση είναι ένα καθοριστικό κριτήριο, δεν είναι όμως και το μόνο που θα αφορά στο στρατηγικό ταμείο αυτό. Θα πρέπει να μπορεί κανένα να διασφαλίσει την επιτυχία των στόχων και αυτό εξασφαλίζοντας ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν τεχνογνωσία για όλους τους ε, τομεί με τους οποίους ε, θα ασχοληθεί το Ταμείο. Βεβαίω υπάρχει ένας κινδύνος πολιτικών στόχων, αυτός όμως πρέπει να εξαλειφθεί. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι ένα τμήμα αυτού του Ταμείου θα χρηματοδοτείται από την αναδιοχέτευση των 3,3 δις ευρώ από το μέσο Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, ε, που αφορούν στον προπολογισμό του 2017 και του 2018. Αρχικά ε, σκοπεύαμε να αυξήσουμε ε, και την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή, τη Γυροπιάνα, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα για να υπάρχει ένα δίκτυο μουσείων και αρχείων. Αυτό το πρόγραμμα το Γυροπιάνα χρηματοδοτείται τώρα από την αναφερθήσα ε, γραμμή του προπολογισμού και δεν θέλω επουδενή αυτό το πρόγραμμα το Γυροπιάνα να απειληθεί από δημοσιονομικές περικοπές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η δική μας Επιτροπή περιορίστηκαν στο να καταθέσουν τροπολογίες στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους. Δεν έχουμε καταθέσει πάρα πολλές, αλλά είναι όλες εξίσου σημαντικές. Με πολύ μεγάλη μου χαρά θα ακούσω τις απόψεις, ελπίζω να με στηρίξετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ, ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Θέλω απλά να σας υπενθυμίσω ότι στις 9.45 θα έχουμε κοντά μας ε, την Επίτροπο Τάισεν. Ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε κλείσει τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Αλλιώς θα προχωρήσουμε μετά τη συζήτηση με την κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία που μας υπέβαλε μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο εισηγητή όταν λέει ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να ενσωματωθεί σε αυτές τις επενδύσεις, σε αυτό το σχέδιο επενδύσεων και το θέμα της καινοτομία στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα για να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη. Είναι μία από τις προτεραιότητες ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ο πολιτισμός θα πρέπει να συμμετάσχουν και να πάρουν ένα τμήμα αυτών των επενδύσεων Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως ασαφείς και γενικές και θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα όσον αφορά αυτό το σχέδιο των επενδύσεων. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για νέα χρήματα τα οποία θα ενσωματωθούν ε, σε αυτές τις επενδύσεις. Οκτώ δις ήδη ουσιαστικά προέρχονται από τον ήδη εγκεκριμένο ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό Connecting Europe Facility, παραδείγματο χάρη, αλλά και άλλα μεγάλα ε, ερευνητικά προγράμματα με ορίζοντα 2020. Θα πρέπει λοιπόν με συγκεκριμένο τρόπο να πούμε και να απαιτήσουμε να μην γίνει εδώ ένα γενικό πρόγραμμα στο οποίο θα ενσωματωθούν χρήματα τα οποία με δυσκολία πετύχαμε να διατεθούν για αυτό το τομέα του πολιτισμού και ξέρουμε ότι όλα αυτά τα προγράμματα, τα ερευνητικά με ορίζοντα του 2020 προέβλεπαν κάποια κονδύλια για τον πολιτισμό. Δεν μπορεί λοιπόν να περιοριστούμε σε αυτά. Το πρόγραμμα αυτό το ερευνητικό είναι ένα από τα σημαντικότερα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολιτισμό και η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να υπάρξουν και άλλα κονδύλια. Πολεμάμε δύο χρόνια με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να διατεθούν αυτά τα κονδύλια σε αυτό το τομέα. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα ξαφνικά αυτά αυτές οι δαπάνες που έπρεπε και είχαν προβλεφθεί να διατεθούν για ερευνητικά προγράμματα ξαφνικά να μεταφερθούν στον τομέα αυτό παρουσιαζόμενα σαν νέα κονδύλια. Η επιστήμη, η έρευνα δεν μπορεί να χάσουν εδώ επενδύσεις και κονδύλια για να μεταφερθούν κάπου αλλού. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό και να προβλεφθούν επιπλέον κονδύλια για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό και επαναλαμβάνω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν αρκεί να ονομάσουν κάποιους τομείς, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες, να πάψουν να είναι γενικές και ασαφείς για να δούμε στην πράξη αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων τι προτίθεται να διαθέσει για τον τομέα του πολιτισμού με αποτελεσματικότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ Πέτρα, ε, Γλέζος τώρα και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν ζήσει το λόγο και κανείς άλλος κλείνει εδώ ερωτώνες. Παρακαλώ κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο. Αγαπητοί Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θεωρώ ότι είναι κάπως πολύ λόγο το θέμα της, ε, των ποσών που πρέπει να δοθούν για το τεράστιο αυτό πρόβλημα που αφορά τις ε, στρατηγικές επενδύσεις πρέπει να ξεκαθαριστεί απολύτως τι ποσό θα δώσουμε για τους αρχαιολογικούς χώρους, τι ποσά θα δώσουμε για τα μουσεία, τι ποσά θα δώσουμε για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που ενασχολούνται με το θέμα, τι ποσά θα δώσουμε για τους ξεναγούς, τι ποσά θα δώσουμε για τη διατήρηση των εθήμων όπως είχε καθιερωθεί η πολιτιστική πρωτεύουσα και όπως προτείνω όχι μονάχα πρωτεύουσα αλλά χωριό κάθε χρόνο από σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ένα χωριό να παρουσιάζει τον πολιτισμό του. Και θα μου πείτε είναι δυνατόν ένα χωριό να έχει πολιτισμό. Το δικό μου το χωριό, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, με 1200 μονάχα κατοίκους έχει πέντε μουσεία και υποίδρυση άλλα τρία μουσεία και έχει και τρεις βιβλιοθήκες. Σας προσκαλώ λοιπόν ιδιαίτερα μια ειδική αποστολή για όποιον αμφιβάλλει από την ε, Επιτροπή μας να επισκεφθεί το χωριό μου για να δει στην πράξη τι σημαίνει πολιτισμός. Και με την ευκαιρία ξανατονίζω αυτό που είπα και στην αρχή της ομιλίας μου. Ο ελληνικός λαός ψήφισε για μια αλλαγή στην πορεία της λιτότητας, της φτώχειας, της ε, μετανάστευσης, της ανεργίας. Μην τον εμποδίζομαι να πάρει πίσω την ψήφο του. Βασικό στοιχείο πολιτισμού είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα ο σεβασμός της θέλησης ενός λαού. Όσοι σκέφτονται και όσοι υπολογίζουν ότι μπορούν να τον εμποδίσουν να ανακτήσει την εθνική του ανεξαρτησία <coughs> και να βγάλει το βρόχο που του έχουν φορέσει οι δανειστές του θα, <coughs> σπάσει τα μούτρα του και καλό <coughs> καλό συγγνώμη όλους τους συναδέλφους με σεβασμό στον πολιτισμό της Ελλάδας με σεβασμό στην ιστορία της Ελλάδας να βοηθήσουν, απευθύνω και πάλι έκκληση, να βοηθήσουν να μην εμποδιστεί ο ελληνικός λαός από την πορεία την οποία χάραξε πριν ένα μήνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Σντρογεύσκη και δεύτερον θέλω να πω το εξής. Ε, δεν θέλω να ε, επαναλαμβάνω, αλλά ξέρετε υπάρχει ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Μιλάμε για 6 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το μόνο ποσό το οποίο δεν προέρχεται από έκτακτα κονδύλια. Όλα τα άλλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτά τα 6 δις προέρχονται από δύο γραμμές του προεπλογισμού. Πρώτον, από τη γραμμή για το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, και δεύτερον από τη γραμμή CEF. E Αν δούμε τώρα από ποιες γραμμές προτίθεται να πάρει η Κομισιόν τα κονδυλιά θα διαπιστώσουμε 2,7 από το πρόγραμμα Horizon 2020, περίπου 2 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας που ασκεί έρευνα σε ε, ε, καινοτομία, τεχνολογία και νεοτερισμούς. Πρόκειται λοιπόν για αυτά που εμάς μας ενδιαφέρουν, δηλαδή να συνδέσουμε την έρευνα με την εκπαίδευση και τις τεχνολογικές εφαρμογές. Και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Είναι δηλαδή ε, σαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απλά να ρίχνει ένα δόλωμα στη θάλασσα και να δει τι ψάρια θα πιάσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πολύ ωραία πείσουμε, λέει η πρόεδρος, η Κομισιόν να δει από πού αλλού μπορεί να πάρει αυτά τα κονδύλια. Η κυρία Τρούπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Να υπογραμμίσω ότι με αυτά τα στρατηγικά σχέδια επενδύσεων θέλουμε να επενδυθούν περισσότερα χρήματα στην κατάρτιση και φυσικά και στην εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας και όλη τη διάρκεια της ε, ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρουμε, και αυτό το συζητήσαμε και στις πρόσφατες μας ανταλλαγές απόψεων, ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην κατάρτιση και να συνεισφέρουν και σε αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων. Είναι και δικό μας βεβαίως καθήκον να πιέσουμε στα κράτη-μέλη μας, ο καθένας το δικό του, να συνεισφέρουν και να παίξουν ε, ε, με τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θα πρέπει να υποβάλει πιστικά προγράμματα, αυτά που θα προσελκύσουν τους επενδυτές, γιατί μόνο έτσι θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο επενδύσεων και θα πρέπει εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην αποσύρουμε κονδύλια από το Horizon 2020, αλλά να υπάρξουν κονδύλια τα οποία θα στοχεύουν και θα επενδυθούν στον τομέα του πολιτισμού και της ε, εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο Σύντροβα. Πρόεδρε, εν πάση εγώ ε, θα ήθελα να στηρίξω τις τροπολογίες του συναδέλφου Σντρογεύσκη. Και θέλω να σας επισημάνω ότι ε, είμαστε σε φάση προετοιμασίας αυτού του ταμείου, αλλά δεν θα πρέπει να μιλάμε για στρατηγικό ταμείο, γιατί αν ήταν στρατηγικό ταμείο θα έπρεπε να προβλέπονται και επενδύσεις ε, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό Όταν όμως εδώ πρόκειται για απόσβεση κονδυλίων, καταλαβαίνετε ότι στον τομέα των επενδύσεων, στον τομέα του πολιτισμού τουλάχιστον, μιλάμε για μακροχρόνιες επενδύσεις. Εκεί στον πολιτισμό δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση ε, γρήγορης, γρήγορων αποσβέσεων των κεφαλαίων. Και επίσης Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην έρευνα και την τεχνολογία η απόσβεση των κεφαλαίων ε, προκύπτει πολύ πιο γρήγορα από ότι στον ε, πολιτισμό. Και γι' αυτό αυτές οι επενδύσεις είναι πιο ελκυστικές για τους επενδυτές. Ε, εμένα με εκπλήσει το ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, αλλά το στρατηγικό ταμείο δεν προβλέπει κονδύλια για αυτό τον τομέα. Δεν προβλέπονται επενδύσεις για τον πολιτισμό. Ε, όπως σας είπα, οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν μακροπρόθεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα στηρίξω αυτή την πρόταση. Ο κύριος Γραμματικάκης έχει το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος ε, κυρία Πρόεδρε, ως συνήθως. Έχω παρατηρήσει το διάστημα που είμαι εδώ ότι ο λόγος, η απόσταση μεταξύ των μεγάλων λόγων του πολιτισμού, του διαφωτισμού που είναι τα θεμέλια της Ευρώπης και της πράξεως είναι πολύ μεγάλη αυτή η απόσταση. Και αντί να μικραίνει από ό,τι φαίνεται και από ό,τι περιγράφηκε από τους προηγούμενους ομιλητές ε, μεγαλώνει. Και νομίζω η αντίδρασή μας σαν Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να είναι εξίσου ισχυρή. Ήδη υπόθηκε από τους ε, συναδέλφους και εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να πω ότι στηρίζω κάθε τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Eh, Σύμφωνο απόλυτα μαζί σας, συνάδελφος Βέρτς, παρακαλώ αν έχετε καλοσύνη και λίγο σύντομα, να είστε σύντομος. Πρόεδρε. Η απασχόληση των νέων είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και υπάρχουν στατιστικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Εδώ και πέντε χρόνια το ποσοστό ανεργίας παραμένει αμετάκλητο, ε, παραμένει παράλλαχτο ανάμεσα στους νέους, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το στρατηγικό σχέδιο του Juncker μπορεί να αποτελεί μια ευκαιρία για να βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσον θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να ε, μειώσουμε την ανεργία των νέων. Γιατί υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και άλλα ταμεία ε, που μπορούμε να συνδέσουμε τα κονδύλια τους με τα κονδύλια του Γιούνκερ για να μειωθεί η ανεργία των νέων και για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσής τους. Δεν ξέρω τώρα μήπως η Επιτροπή επιθυμεί να προσθέσει κάτι άλλο γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει τα μάλα η ενεργός συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι θα υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της εκπαίδευσης. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε εσείς να μιλήσετε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήδη αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι πολύ θετικό για τον τομέα του πολιτισμού και περιέχει πολλά στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την καινοτομία και για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Θεωρώ πραγματικά ότι ο δημιουργικός τομέας ε, θα πρέπει φυσικά και να στηριχθεί, προβλέπεται αυτό από το σχέδιο επενδύσεων, στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιος μίλησε επίσης και για τις υποδομές των αστικών περιοχών, για αθλητικές, παραδείγματος χάρη, εγκαταστάσεις ή για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο έχει σαν σκοπό να γίνει η επιτυχής μόχλευση ιδιωτικών κονδυλίων. Και φυσικά σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές που θα επιτρέψουν σε αυτά τα έργα να χρηματοδοτηθούν από δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια. Πράγματι λοιπόν αυτή είναι η πρόκληση και ελπίζω να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και με τη δική σας βοήθεια. Ε, τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο που είναι κοντά μας. Μόνο αν έχει την καλοσύνη ένα λεπτό κύριε Επίτροπο, υπομονή για να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που δείξατε. Θα προσπαθήσω όσον αφορά τις τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 5, να ενισχύσω τους στόχους ε, όπως αναφέρθηκαν έτσι ώστε ο ψηφιακός κόσμος, ο κόσμος του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, όλες αυτές οι καινοτόμες και δημιουργικές ε, προσπάθειες να στηριχθούν. Έχω και μια τελευταία παρατήρηση. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, δεν πρέπει να είμαστε ακραίοι και υπερβολικοί, γιατί αλλιώς θα απορριφθούν οι τροπολογίες μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι πέρα από την ουσία να προωθήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα με πολιτιστικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ε, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Έκων και Μπάτς μας έχουν ε, εξηγήσει τις απόψεις τους. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι να εκφράσουμε την απόψή μας με απόλυτη αποφασιστικότητα στην Ολομέλεια. Και νομίζω ότι η δική μας η Επιτροπή θα συμμετέχει περισσότερο με σκιώδεις ηγητές, ε, θα συμμετέχουμε δηλαδή στα σημεία εκείνα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρουν ε, στο τομέα των αποφάσεων. Άρα δηλαδή, ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το να φαινόμαστε, αλλά με ενδιαφέρει η ουσία των επιχειρημάτων και επίσης ε, και το ότι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση θα πρέπει να καταλαμβάνουν μεγαλύτερη θέση. Υπάρχουν πέντε προτεραιότητες, υπάρχει η εκπαίδευση, αλλά δεν υπάρχει τόσο όσο η δημιουργικότητα, ο δημιουργικός πολιτισμός. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη Λετωνική Προεδρία. Τώρα θα ήθελα ε, να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δείξατε έτσι υπομονή ε, και Νομίζω ότι συναντήκαμε την 1η Οκτωβρίου, τότε δηλαδή που ήταν η ακρόαση από κοινού με την Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Ε, αυτό το χαρτοφυλάκι που πήρατε είναι καθοριστική σημασία για μας και μεταξύ άλλων στις 3 η ώρα το απόγευμα έχουμε κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση των σχολικών συστημάτων, της ε, απασχόλησης των νέων και θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε περίπου κάποια λεπτά, καμιά δεκαριά και μετά θα δούμε τι είδου ε, ερωτήσεις υπάρχουν, θα τις ομαδοποιήσουμε για να υπάρξει και ένας δεύτερος ε, γύρος ε, απαντήσεων από εσά και στο τέλος πάλι θα συνεχίσουμε. να σας πω το εξής, ευθύς εξ αρχής. Το πρώτο, ότι η Επιτροπή Πολιτισμού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει μια σφαιρική αρμοδιότητα για θέματα ε, παιδείας, παρότι στην Επιτροπή έχουν ε, μετατεθεί λιγάκι τα ε, θέματα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και των προσόντων. Αυτά πήγανε στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει η διαβίου μάθηση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε Υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δεν θέλουμε να χαθεί. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι είδους μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλιστεί όχι μόνο η σταδιακή ε, μετάβαση αλλά και η σχέση που θα έχουμε με τη Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης η δική μας Γενική Διεύθυνση με αυτήν της Απασχόλησης κάτι άλλο Θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη δική σας τη θέση σε σχέση με τις νέες στρατηγικές ε, και πολιτικές ε, που έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται όσον αφορά τους μηχανισμούς εγγύησης για τους νέους, ε, την συνεργασία με τομείς που έχουν σχέση με τη γνώση. Με την συνάλφο Λιμπάτσκα έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση που αφορά στη διαδικασία της Μπολόνια και μία άλλη έκθεση τα αφορά ε, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Για να δείτε λιγάκι σε τι θέματα έχουμε ήδη ξεκινήσει τι εργασίε μας. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η ευρύτερη συνεργασία σε όλου αυτού του τομεί. Αυτό όμω που μα απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μία ολιστική προσέγγιση ε, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές προκλήσεις υπό την προπόθεση τη ευφυούς ανάπτυξη, όπω αναφέρεται. Δηλαδή όχι έτσι στιγνές πολιτικές, αλλά έτσι κάποια ευρύτερη λογική. Εμάς αυτό μας απασχολεί όλα αυτά κάτω από αυτό το πρίσμα που σας παρουσίασα και περιμένουμε τη δική σας την άποψη. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που επανέρχομαι εκεί από όπου ξεκίνησα. Βλέπω πολλά καινούργια πρόσωπα και ελπίζω η προσωπική σας ζωή να είναι εξίσου ευτυχής με τη ζωή σας στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας ε, μία εισαγωγή, θα την κάνω στα αγγλικά. Είμαι βεβαίω στη διάθεσή σας μετά για ερωτήσεις. Επειδή έχουμε και τους διερμηνείς μας θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα μετά, στα Ολλανδικά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω ως Επίτροπος Αρμόδια για τις κοινωνικές υποθέσεις, την απασχόληση, την κινητικότητα και τις δεξιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με μια θετική νότα. Θα ήθελα να πω ότι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας υπήρξαν πηγή ε, ε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Στο τέλος του 2014, 500.000 λιγότερα άτομα ήταν άνεργα από ό,τι το προηγούμενο χρόνο και προβλέπουμε ότι η ανεργία θα συνεχίσει την πτωτική της τάση το 2015 και, και πιστεύουμε ότι πραγματικά το έχω είναι κάτω από το 10% γιατί ε, αυτό είναι που το οποίο καταλήξαμε το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ας μην ε, πανηγυρίζουμε όμως και ας μην είμαστε αυτάρεσκοι γιατί έχουμε ακόμα 24 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη που δεν έχουν εργασία, που είναι άνεργα και γνωρίζουμε ότι μεταξύ αυτών των ανθρώπων συμπεριλαμβάνονται 5 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι, δηλαδή από 15 ως 24 άνθρωποι νέοι που είναι άνεργοι και ξέρουμε ότι το 33% εξ αυτών είναι άνεργοι για πάνω από ένα χρόνο και κατατάσσονται στην κατηγορία των ε, ε, ε, άνεργων μακράς δικασίας. Λοιπόν, το βασικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως για τα 5-7 εκατομμύρια νέων που είναι άνεργη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, που δεν θα προκύψουν ε, από ένα μαγικό κόλπο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια και θα πρέπει να κάνουμε σωστές και έξυπνες επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω δύο λόγια σχετικά με το πακέτο επενδύσεων το πρόγραμμα επενδύσεων που προετάθη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Το ονομάζουμε σχέδιο Juncker στην Επιτροπή. Αυτό δεν είναι μόνο ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Πώς θα το έλεγα, είναι ένας νέος πυλώνας στο τρίγωνο, το οποίο θα στηριχθεί η νέα αυτή η Επιτροπή Juncker θα συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στο θέμα των, ε, του προπολογισμού, στο θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελούσε μέρος των στόχων της προηγούμενης Επιτροπής, αλλά θέλουμε να προσθέσουμε και κάτι γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με φορολογική υπευθυνότητα και μόνο με την δημοσιονομική σταθερότητα και τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, αλλά γνωρίζουμε ότι απαιτούνται επενδύσεις. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν κρατικά κονδύλια για όλες τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν χρήματα ενυπνώσει και θα πρέπει πολλά από αυτά να τα επενδύσουμε, να τα διοχετεύσουμε στην αγορά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα, για τα κονδύλια, για να δώσουμε εγγυήσει στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσει να προσελκύσει κονδύλια σε επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη ποιότητα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος εργασίας αυτής της νέας επιτροπής. Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε εμείς είναι όταν υπάρχουν οι νέες αυτές ευκαιρίες να υπάρχουν οι άνθρωποι που θα τις αδράξουν. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επενδύσουμε στις δεξιότητες, στις γνώσεις, ιδιαίτερα για τους νέους και για τους μακροχρόνια άνεργους, αλλά και για όλους τους άλλους, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί η διαβίου μάθηση στην εποχή μας είναι κάτι αναγκαίο. Έχουμε προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κάνουν αυτό, επενδύουν πάνω από 80 δισεκατομμύρια, νομίζω ότι είναι 86 δισεκατομμύρια. Επενδύουμε λοιπόν 86 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 7 χρόνια. Η πρότασή μου να προωθήσουμε την προχρηματοδότηση μέσω της ε, πρωτοβουλίας με ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι κάτι που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου φέτος και έχει σκοπό, Πω να βοηθήσει 650.000 περίπου νέους ανθρώπους έτσι ώστε να ενταχθούν το συντομότερο στην αγορά. Ζητήσαμε από τις χώρες μέλη να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τους νέους, αλλά πολλές χώρες, σε πολλές χώρες μέλη δεν οι ρυθμοί δεν είναι αρκετά ε, γοργοί, υπάρχουν ε, περιορισμοί και δεν υπάρχουν χρήματα, επαρκή κονδύλια για χρηματοδότηση. Κάναμε κάτι εξαίρεση το σύστημα των διαθροτικών ταμείων, δώσαμε μία προχρηματοδότηση κατά 30% από την αρχή κιόλας και πιστεύουμε ότι αυτό δείχνει το πόσο έχει δεσμευτεί η Επιτροπή αυτή στο να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο τους νέους. Και πιστεύω ότι όλοι συμφωνείτε με αυτή τη δέσμευση. Παράλληλα έχουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να διασφαλίσουν ε, ανάπτυξη και ένα φιλικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, απλοποίηση των φόρων, καλύτερη διασύνδεση των συστημάτων κατάρτισης, ε, εκπαίδευσης και την ε, αγορά εργασίας. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να παράσκουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για μεγαλύτερη απασχολησιμότητα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη κατανόηση και να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των ετούντων ε, απασχόλης και των εργοδοτών. Αυτό βεβαίως δεν ε, σημαίνει την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών του α ή β εργοδότη. Σημαίνει ότι θα πρέπει να προλάβουμε, να διαγνώσουμε των προτέρων τις τάσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν καλύτερη, μεγαλύτερη δυνατότητα να απασχοληθούν σε μία θέση εργασίας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη σταδιοδρομία του κάθε ανθρώπου. Βεβαίως θα χρειαστούν νέες δεξιότητες, ξέρουμε ότι επέρχονται γοριές αλλαγές στην τεχνολογία, στη ζωή και αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις αυριανές εργασίες δεν τις έχουμε ακόμα φανταστεί. Ξέρουμε ότι η υψηλή ανεργία συνηθίζει υπάρχει με έλλειψη δεξιοτήτων σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. Και υπάρχουν δύο είδη αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Καταρχάς έλλειψη δεξιοτήτων για τις οποίες υπάρχει, αίτηση, ε, υπάρχει ζήτηση και έχουν σχέση με την καινοτομία και από την άλλη έχουμε περιορισμένη απασχόληση, δηλαδή υπάρχουν άτομα που δέχονται εργασίες ε, για τις οποίες τα προσόντα τους είναι περισσότερα από αυτά που χρειάζονται <clears throat> και αυτό το κάνουν γιατί δεν βρίσκουν την κατάλληλη εργασία. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων θα μπορούσαν να έχουν ε, σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ποιες είναι, για ποιες ε, δεξιότητες υπάρχει ζήτηση πέρα από τις ειδικότητε και ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες μέλη υπάρχει έλλειψη ορισμένων δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την ε, πληροφορική, με την τεχνολογία. Ξέρουμε όμως παράλληλα ότι χρειαζόμαστε και άλλες δεξιότητες. Χρειαζόμαστε επιχειρηματικές δεξιότητες ε, από πλευράς ανθρώπων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, αλλά χρειαζόμαστε και ανθρώπους ικανούς να μετατρέψουν την ιδέα σε πράξη. Ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν ορισμένα προγράμματα. Γλωσσικές ικανότητες, ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα είναι ε, θέματα που απασχολούν τους εργοδότες και βεβαίως οι κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει επίσης ε, να έχουν τη δέουσα προσοχή. Η σχετική πείρα βεβαίως αυξάνει τις πιθανότητες απασχολησιμότητας. Ε, πήρα Κάτι που αφορά και τους νέους ανθρώπους. Αυτό μπορούν να το κατακτήσουν μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που συμπεριλαμβάνουν και εργασία ή μαθητεία ή διτή, ε, το διτό σύστημα. Αυτό μπορεί να δώσει στους μαθητευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα όσα έχουν μάθει. χωρίς με ισχυρά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας έχουν καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την απασχολησιμότητα των νέων συμπεριλαμβάνοντας και μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως τα άτομα που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο ή άτομα που δεν ε, ασχολούνται ούτε με την κατάρτιση ούτε βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Αυτό που επίσης μετράει είναι κατά πόσον υπάρχει κάποιος σεβασμός από πλευράς της κοινωνίας, των γονιών και των μαθητών σε ό,τι αφορά την μαθητεία και την κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να είναι μία πρώτη επιλογή και όχι μία δεύτερη επιλογή. Το να ανοίξουμε την πόρτα, γιατί ε, ανοίγει την πόρτα σε καλές εργασίες. Γι' αυτό στη διαδικασία της Κοπεχάγης στην επόμενη φάση θα ήθελα να δώσω προτεραιότητα σε αυτό που μπορεί να κάνει η Επιτροπή για να υποστηρίξει στηρίξει τις χώρες μέλη για να εξυγχρονίσουν τα συστήματά τους και να αυξήσουν ε, να ενισχύσουν την επαγγελματική κατάρτιση. Είμαι επίση πεπισμένη ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερου παίκτε, συμπεριλαμβάνοντα και μικρομεσαίε επιχειρήσει, έτσι ώστε να αυξήσουν την παροχή, την ποιότητα και την γενική εικόνα που προβάλλεται σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντα και μία ενδυνάμωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μαθητεία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερε ευκαιρίε για του νέου για να μπορέσουν να απασχοληθούν γιατί περί αυτού πρόκειται. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως υπάρχει για το θέμα της μάθησης των ενηλίκων. Είναι σημαντική η πρώτη εργασία, αλλά είναι επίσης σημαντικό το να μπορεί κανείς να παραμείνει σε μία δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη διαβίου μάθηση. Υπάρχουν ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν τα πετούμενα προσόντα. Κάνουν μια χαμηλά αμεβόμενη δουλειά που δεν τους δίνει την δυνατότητα να αναζητήσουν κάτι καλύτερο γιατί τους λείπουν οι δεξιότητες. Θα μπορούσαν ε, λοιπόν αυτοί να, είναι ε, να, να χρησιμοποιήσουν ένα εφαλτήρα για να προχωρήσουν. Πολιτικές που αφορούν τις δεξιότητες. Ε, είμαι πεπισμένη ότι παίζουν ζωτικό ρόλο στην αγορά εργασίας. Το δικό μου χαρτοφυλάκιο δείχνει τη σημασία που αποδίδεται σε μια καλύτερη ευθυγράμμιση, καλύτερο ε, καλύτερη αντιστοίχηση δεξιοτήτων και εργασίας. Βεβαίως οι δεξιότητες δεν αναπτύσσονται σε ένα κενό, αποτελούν ένα προϊόν εκπαίδευσης και εμπειρίες. Μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι θα συνεργαστούμε στενά με τον Πίτρο Ποναβράτσι για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει ένας παραλληλισμός ε, εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω σήμερα, αλλά όχι μόνο σήμερα, και στο μέλλον σχετικά με το πώς θα έχουμε την βεβαιότητα ότι θα μπορούσαν οι δεξιότητες των λαών να διαμορφώσουν το μέλλον. Η κοινωνική αγορά της Ευρώπης θα πρέπει να δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα για μια αξιοπρεπή και καλά αμοιβόμενη εργασία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας για μια ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Επίτροπο Τάισεν για την σαφέστατη παρέμβασή της, αλλά και γιατί, για την τοποθέτησή της. Ήταν σαφές ότι υπάρχει διάθεση στενής συνεργασίας Σήμερα στη συνάντηση των συντονιστών θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και για αυτή την προκαταβολή του 30% αυτό είναι κάτι που ζητήθηκε και από το Κοινοβούλιο και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η απόφαση που πήρατε καθώς και η προσέγγιση που ακολουθήσατε που δείχνει ότι έχετε απόλυτη κατανόηση αυτού του θέματος και της ανάγκης να υπάρχει, ε, να εστιάσετε την προσοχή σας προς την διαβίου μάθηση. Υπάρχει πραγματικά ανάγκη να υπάρξει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας προβλέποντας τις νέες μορφές ε, εξειδικεύσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας αυτός που βρίσκεται εκτός τώρα. Θαυμάσια βάση εργασίας. Τώρα, να δούμε ποιοι είναι οι εγγεγραμμένοι για να πάρουν το λόγο. Ήδη, α, ήδη μαζεύονται πολύ. Ωραία. Κιούτσοκ, Τρούπερ, Βέρντ, Γραμματικά, Σφεράιαν, Μπάτσκα, Νέκοφ, Σεντρόβα και Μόργανο. Κιούτσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας κίνησης και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άξα αυτά που είπατε, αλλά δεν ήταν ε, σαφές ε, όσον αφορά τις δράσεις που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί παρόλο που υπάρχει πολύ σημαντική ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές κενές θέσεις στην αγορά εργασίας σε κάποιες χώρες, νομίζουμε ότι δεν γίνονται αρκετά έτσι ώστε μία από τις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε, ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία κίνησης και κυκλοφορίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Μήπως να συγκεντρώσουμε περισσότερες ερωτήσεις για να απαντήσετε ομαδικά. Ε, κυρία Τροπολή, ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπο για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση, διαβίου μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και βεβαίως αυτά σε σχέση με την οικολογική μετάβαση η οποία είναι απαραίτητη. Μιλάτε για νέες δεξιότητες, μιλάτε για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων έτσι ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς αυτή να συνοδεύεται απαραίτητα με μια αύξηση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Πώς προτίθεστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Χρειάζονται έξυπνες επενδύσεις, καθότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε από την ανάπτυξη ε, το θέμα αυτό της οικολογικής μετάβασης. Ευχαριστώ πολύ. Η Julie Ward έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εγώ, όσον αφορά την αισιοδοξία, την προσεκτική αισιοδοξία που εκφράζεται, μπορώ να πω ότι έχω πολλές αμφιβολίες. Βλέπω μεγάλη απόγνωση στην εκλογική μου περιφέρεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι είδου θέσεις απασχόλησης σκέφτεστε, γιατί βλέπουμε πραγματικά όλο και περισσότερους άνεργους νέους να ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Επίσης εργαζόμενους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Έχουμε μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων, νέων Ευρωπαίων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουμε αποτύχει. Σήμερα πρέπει να δώσουμε ελπίδα στους νέους της Ευρώπης, να τους δώσουμε κάποιες προοπτικές για το μέλλον. Δεν πρόκειται για εργασία που να μοιάζει με τη σκλαβιά. Οι δικές μας παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι προς όφελος αυτής της νέας γενιάς. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούνται τα προσόντα τους, η δημιουργικότητά τους, τα ταλέντα τους, ότι μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία μας, ότι τους επιτρέπουμε να είναι δραστήριοι και ενεργά μέλη της οικονομικής μας ε, κοινότητας στην Ευρώπη και να μπορούν να βρουν θέσεις απασχόλησης που να τους ανταμείβουν. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρωτοβουλίες της. Θα πρέπει να λάβει υπόψη στην κοινωνική πτυχή, την πτυχή της απασχόλησης. συνεργασία λοιπόν με άλλες επιτροπές, η δική μας επιτροπή ασχολείται με αυτά τα θέματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιες άλλες επιτροπές που στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην ανάπτυξη, στην οικονομική πτυχή, δεν παίρνουν καθόλου σοβαρά υπόψη όλη αυτή τη χαμένη γενιά των νέων στην Ευρώπη. Οι νέοι της Ευρώπης, κατά την άποψή μας, είναι σημαντικοί εταίροι αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς. Και βλέπουμε νέους να έρχονται εδώ, στην Επιτροπή μας, στις εργασίες μας, με έμπνευση, με όρεξη για δουλειά, με δεξιότητες και με ταλέντα. Είναι όμως σαν να μην τους αντιμετωπίζουμε σαν έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς αυτής της προσπάθειας, σαν ενδιαφερόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γραμματικάκης έχει το λόγο. Νομίζω, κυρία Πρόεδρος και η κυρία Κομίσιονερ, ότι είναι σημαντική η σημερινή μέρα και συγχαίρω και τους δύο για την οργάνωσή της. Θα μιλήσω πολύ γρήγορα σαν καθηγητής θα μιλήσω μετά σαν Ευρωβουλευτής και το συμπέρασμα. Κρίνοντας σαν καθηγητής στην ομιλία της κυρίας ε, Κομίσιονερ ήταν εξαίρετη. Είχε επιχειρήματα, είχε δομή και είχε και άποψη. Ε, σαν Ευρωβουλευτής όμως πηγαίνω εδώ στον πίνακα που μας είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε και βλέπω ότι το unemployment, το rate of unemployment είναι ας πούμε στη χώρα μου 58% στην Ιταλία 40% στην Ισπανία 55% και ούτω καθεξής εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι οι προσπάθειες της Κομισιόν είναι μεγάλες, δύσκολες και θα έλεγα επίμονες. Όταν όμως κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή η εξαίρετη θεωρία δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, η θεωρία αυτή τη στιγμή και η πραγματικότητα είναι τα στοιχεία που μας παραθέτεται, κάτι δεν πάει καλά με τη θεωρία. Και θα κλείσω, είμαι πάντα σύντομος όπως ξέρετε, ε, φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τα μαύρα θα μεγαλώνουν στις χώρες και θα έχουμε στο τέλος μια μαύρη Ευρώπη, μια απεγνωσμένη Ευρώπη, πράγμα που κανείς δεν το επιθυμεί, άρα πρέπει να αλλάξουμε τη θεωρία. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να την αλλάξουμε, ίσως να πάυσουμε λίγο τη λιτότητα, ίσως να σκεφτούμε άλλους τρόπους, αλλά είναι επίγον, επαναλαμβάνω, ως καθηγητής, ως ευρωβουλευτής και ως φίλο Ευρωπαίος, να αλλάξουμε τη θεωρία. Ευχαριστώ πολύ. Φεράιαν, καταρχήν να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσίασή της και για το ότι προτείνει συνεργασία μεταξύ ημών γιατί πρέπει να στηρίξουμε τον τομέα του πολιτισμού. Το βεβαίως ε, βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες τα, τα συστήματα, τα εκπαιδευτικά, επαγγελματική κατάρτιση με την καθαρά ακαδημαϊκή σχολική εκπαίδευση έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την στήριξη αυτών των συστημάτων στις χώρες που το προτείνουν και θέλουν να τα ενισχύσουν. Δηλαδή, συνεργασία μέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ της μαθητείας, συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και του καθαρά σχολικού θεωρητικού συστήματος προτίθεστε να στηρίξετε αυτές τις δομές, αυτές τις ε, προσπάθειες, αυτές τις πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το γιατί σε κάποιες χώρες τα συστήματα αυτά έχουν καλά αποτελέσματα και τη λειτουργούν αποτελεσματικά και σε άλλα όχι. Και μήπως πρέπει να δούμε πού αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε περισσότερο, να στηρίξουμε την επαγγελματική κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί βλέπουμε τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται ίσως καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη πληροφόρηση, πώς βελτιώνονται οι ικανότητες μάθησης και τα συστήματα αυτά, πώς τα κάνουμε λίγο πιο αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δεσμευθούμε και να επενδύσουμε εκεί που υπάρχει αποτέλεσμα. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει και μια καλή ε, ένα καλό προγραμματισμό γιατί σκοπός μας είναι τα αποτελεσματικά αυτά συστήματα να οδηγήσουν σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τους νέους της Ευρώπης. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική εδώ και η κινητικότητα, η προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των νέων εκεί που υπάρχουν και διαπιστώνονται περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σήμερα κινήματα μετανάστευσης των νέων για να μπορέσουν να ενσωματωθούν σε κάποια άλλη αγορά εργασίας, αλλά Βλέπουμε επίσης ότι χρειάζεται και κάποια προσαρμογή. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιστροπή στηρίζει βεβαίως προγράμματα που βοηθούν τους νέους να ενσωματωθούν σε κάποια άλλη αγορά εργασίας, αλλά ίσως εδώ θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες οι δράσεις. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι τώρα πια έχουν μαζευτεί αρκετά επιχειρήματα και τώρα νομίζω ότι μπορείτε να τα απαντήσετε κι εσείς έτσι συνολικά όλα μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν υπήρξε μια ερώτηση για την κινητικότητα στην Ευρώπη. Τι μπορούμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε. Να σας απαντήσω με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Καταρχήν στηρίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία, την κινητικότητα, είναι ένας από τους πυλώνες των ευρωπαϊκών συνθήκων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στηρίζουμε αυτήν την ε, θεμελιώδη ελευθερία, πάρα πολύ σημαντική για την οικονομία της Ευρώπης ε, και για την ε, στήριξη της κοινωνικής αυτής συνοχής. Υπάρχουν κανόνες λοιπόν στις συνθήκες, υπάρχουν και σημαντικοί τομείς στους οποίους προωθούνται οι προσπάθειες αυτές κινητικότητας. Υπάρχει οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, υπάρχει εξάλλου και η οδηγία αυτή η οποία ψηφίστηκε πέρσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγρυπνεί έτσι ώστε αυτά τα σημεία που εμπεριέχει αυτή η οδηγία να εφαρμόζονται και να τηρούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως το θέμα της κινητικότητας προκαλεί και πολλά ερωτηματικά. 3,3% μόνο των Ευρωπαίων εργαζόμενων μετακινούνται για να εργαστούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Δεν είναι πολύ αυτό το ποσοστό, 3,3%. Πολλοί θεωρούν σήμερα ότι αυτοί οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, αυτοί οι εργαζόμενοι που φεύγουν από τη χώρα τους για να εργαστούν κάπου αλλού, απειλούν την αγορά εργασίας κάποιου άλλου κράτους μέλους. Ότι υπάρχουν καταχρήσεις, ότι εποφελούνται από τα κοινωνικά ωφέλη ενός άλλου συστήματος. Αυτό όμως το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό. Για το 2015 έχουμε εγκρίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λεγόμενο πακέτο για την κινητικότητα. Καταρχήν θέλουμε να κάνουμε τον απολογισμό αυτών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Με στοιχεία, με αριθμούς. Να εξετάσουμε ποιες είναι οι μεσταναστευτικές ροές η λεγόμενη φυγή των εγκεφάλων που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη. Να προσπαθήσουμε λοιπόν με πραγματικά στοιχεία και αριθμούς να, κάνουμε έναν πραγματικό απολογισμό. Και κατόπιν, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, να κάνουμε κάποιες προσωμιώσεις. Να αλλαλήσουμε τα στοιχεία, να δούμε ποιες είναι οι τάσεις για το μέλλον και να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη αυτή η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ποια είναι η πρακτική στα κρατημέλη. Τα κρατημέλη καλούνται εδώ να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία αυτής της οδηγίας στην πράξη. Τι ακριβώς γίνεται λοιπόν. Θα εξετάσουμε επίσης και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν καταχρήσεις. Υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες πού μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση και όσον αφορά τον συντονισμό για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ίσως να χρειαστούν κάποιες αλλαγές, κάποιες μεταρρυθμίσεις. Είναι λεπτό το θέμα και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εδώ να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν. Το πακέτο πάντως αυτό για την κινητικότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το EURES. Επίσης, θέλουμε να το ενισχύσουμε, γιατί σκοπός μας είναι η επαγγελματική κινητικότητα να ενισχυθεί, να πλαισιωθεί και να ενισχυθεί. Και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. 24 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη και βεβαίως σε καμία περίπτωση η κατάσταση αυτή δεν είναι ικανοποιητική. 24 εκατομμύρια άνεργοι, ένας πολύ σημαντικός αριθμός και την ίδια ώρα 2 εκατομμύρια κενές θέσεις. Με την κινητικότητα ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτή την αναντιστοιχία. Στη δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε θα απαντήσω ως εξής. ποιες αλλαγές θέλουμε να υιοθετήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική στήριξη των κρατών μελών. Ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη όπου διαπιστώνουμε δυσκολίες στην αγορά εργασίας ή εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται μεν, δεν μπορούν όμως να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Εργαζόμενου σε κατάσταση φτώχειας δηλαδή. Θα πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν το θέμα της κατάρτισης, της ε, διαβίου κατάρτισης, την εξέλιξη στην αγορά εργασίας και την αναντιστοιχία που σαφώς συνεχίζει και υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Βεβαίως υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, αλλά σαφώς και θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ε, εργαζόμενους. Προσπαθώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου, με συγχωρείτε. Μιλήσατε για την προσεκτική μου ή επιφυλακτική μου αισιοδοξία. Ίσως να φάνηκα πολύ αισιόδοξη. Παρόλα αυτά, όταν παίρνω το λόγο, όταν κάνω μία παρουσίαση και αναφέρω τον αριθμό των μακροχρόνια άνεργων, των νέων άνεργων, βεβαίως αυτοί οι αριθμοί είναι σωστοί, αλλά δεν είναι σωστό να ξεκινάμε πάντα με αυτούς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε μια θετική επίδραση επί αυτών. Έχουμε κονδύλια, έχουμε εργαλεία, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη. Εγώ βλέπω ελπίδα βλέπω μία μικρή ανάκαμψη. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη, χωρίς να είμαι αφελής. Απλώς συνεχίζω να ελπίζω και με ενεργό τρόπο θέλω να βοηθήσω έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η κοινωνία μας το θέμα των νέων τώρα. Έχουμε την εγγύηση για τους νέους, Youth Guarantee, με τη δέσμευση των κρατών μελών που απευθύνεται σε νέους που είτε έχουν εγκαταλείψει πολύ νωρίς το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς κάποιο πτυχίο, είτε νέους άνεργους ε, θέλουμε να τους επαναφέρουμε σε κάποια προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εμπειρία, νέες προοπτικές, να μπορέσουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Βεβαίως Σκοπός μας δεν είναι να τους τοποθετήσουμε κάπου, χωρίς μέλλον, χωρίς εξέλιξη. Γι' αυτό και μίλησα για τα 350 δις του σχεδίου Juncker. Δεν φτάνουν, θέλουμε πολύ περισσότερα. Καταλάβατε ποιο είναι το μήνυμα. Καταλάβατε ποια είναι η ερμηνεία μας όσον αφορά την ρήτρα ευελιξίας του Σύμφωνο Σταθερότητας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ευελιξίες για τις διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Οι μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν ευελιξία, θα δημιουργήσουν περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη με αυτή την ευελιξία να μπορέσουν να φτάσουν πιο εύκολα, δίνοντάς τους λίγο περισσότερο χρόνο στους μεσοπρόθεσμους στόχους τους θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης ποιότητας και βεβαίως όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά που γίνονται με τον ορίζοντα 2020. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εγώ, σαν αρμόδια επίτροπος, Φυσικά και θέλω να ενσωματώσω όλη αυτή τη δράση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό αποτελεί ένα τμήμα της στρατηγικής για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν αρμοδιότητα την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την βελτίωση των δεξιοτήτων, την ισότητα. Και καταρχήν οι δύο λέξεις που θα ήθελα να κρατήσω είναι ανάπτυξη και καταρχήν απασχόληση. Βάζω σαν νούμερο ένα προτεραιότητά μας την απασχόληση πριν από την ανάπτυξη. Και αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, να συντονίσουμε τις δράσεις μας, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμός και αυτό είναι η κύρια, αν θέλετε, ενασχόληση όλων των επιτρόπων. Όλων των επιτρόπων, όχι μόνο η δική μου. Είμαστε όλοι πεπισμένοι, καθώς και ο πρόεδρός μας, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη δράση μας για να ενισχύσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Κύριε Γραμματικάτη, είστε καθηγητής και ευρωβουλευτής. Κι εγώ ήμουν ευρωβουλευτής για πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό και το σέβομαι ιδιαίτερα το επάγγελμα του ακαδημαϊκού. Ένας καλός δάσκαλος πραγματικά μπορεί να κάνει πολλά και σέβομαι ιδιαίτερα αυτό που κάνετε. Νομίζω ότι ενδεχομένως απάντησα εν μέρη στην ερώτησή σας. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε και αν πρέπει να εγκαταλείψουμε την λιτότητα. Η απάντησή μου είναι όχι. Χρειαζόμαστε δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλιώς δεν μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Χρειαζόμαστε τις αγορές. Χρειαζόμαστε τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει και διαρθρωτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αλλά και δημοσιονομική σταθερότητα. Πρέπει να ξυπνήσουμε τις επενδύσεις τον ιδιωτικό τομέα για να επενδυθούν κονδύλια σε νέους τομείς, να δημιουργηθούν ποιοτικέ σχέσεις απασχόλησης. Και βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας για να επενδυθούν κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα εξαρτώνται από τις τράπεζες. Αλλά χρειάζονται και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης πέραν από τις χρηματαγορές. Και τώρα απαντώ στην τελευταία ερώτηση, πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτουργούν με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Ήμουν στο Βερολίνο και επισκέφτηκα την Siemens με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που χρηματοδοτεί η Siemens για τους νέους οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είμαστε παρόντες λοιπόν. Και βεβαίως διαπιστώνουμε ότι μεγάλος αριθμός νέων επιθυμεί να εποφεληθεί από μια τέτοια επαγγελματική κατάρτιση και κάποιους από αυτούς, η μισή περίπου, δεν ολοκληρώνουν αυτή την κατάρτιση. Ξέρουμε σήμερα ότι το 85% αυτών που ολοκληρώνουν ένα τέτοιο σεμινάριο ή πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν κατόπιν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και ενσωματώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις πρωτοβουλίες, να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες προσπάθειες έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα αυτής της ε, κατάρτισης που προτείνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα κάποιων κρατών. Μπορώ να σας στείλω εξάλλου και στην πρόεδρο της Επιτροπής σας όλες τις πρωτοβουλίες τις οποίες ενισχύουμε. Χρειάζεται ένα σύστημα διοικητικό έτσι ώστε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτών των συστημάτων κατάρτισης να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και χρειάζονται και αποτελέσματα σε αυτή την κατάρτιση. Δεν πρέπει απλώς να προτείνουν οι επιχειρήσεις κάποια σεμινάρια. Πρόκειται για την κατάρτιση των νέων μας. Πρέπει να αλλάξουν λοιπόν νοοτροπία οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι από κοινού λοιπόν να αναλάβουν αυτές τις προσπάθειες και δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλοί νέοι επιθυμούν να ενσωματωθούν σε αυτά τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για μία πιο υποβαθμισμένη κατάρτιση. Αυτό είναι πολύ κρίμα γιατί αυτό δημιουργεί μια απογοήτευση στους νέους μας. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν δεξιότητες και ταλέντα στους νέους μας, τις οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Και πρέπει να αναβαθμιστεί η εικόνα αυτών των ε, ε, εναλλακτικών ε, εκπαιδευτικών συστημάτων στα μάτια των γονιών, στα μάτια των είδων των νέων. Έτσι ώστε να είναι μια πραγματική επιλογή. Χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πολλούς τομείς και πρέπει πραγματικά να σεβόμαστε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Παρακαλώ θερμά τους συναδέλφους να είναι λακωνικοί γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχω έναν εκτενή κατάλογο. Συνάρφη, Λιγάς, Ταμέρους, Σορμπόρτα, Αγγλέζος, Χέιχολμ και τελειώνουμε εδώ. Θερμή παράκληση. Ένα λεπτό η ερώτησή σας. Διαφορετικά δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ, εδώ, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, αλλά ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για μία φράση που είπατε. Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό υπέρ της κατάρτιση. Γιατί η δυνατότητα να προβλεφθεί κάποια κατάρτιση, κάποια μαθητεία που είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του διτού συστήματος είναι κάτι που απαιτείται σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, ακόμα και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Το πρόβλημα βέβαια είναι να έχει κανείς τη δυνατότητα να κάνει κάπου αυτή την πρακτική εξάσκηση και να προκύψει για κάποιο πλεονέκτημα. Θα ήθελα λοιπόν στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας να σκεφτείτε ποια θα μπορούσε να ήταν μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφόρησης, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το που μπορεί κανείς να κάνει μια πρακτική εξάσκηση. Βεβαίω, ε, δεν μιλάμε για γίγαντες, για την ε, Volkswagen, ε, για τι ζήμε. Αυτοί δεν μπορούν βεβαίως να εξασφαλίσουν μια θέση σε όλου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι. Συνάδελφο Νέκοφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως ε, τα κονδύλια που έχουν προβλεφτεί για την ε, καταπολέμηση ανεργία των νέων είναι πρόσδεκτα στις αρχές του 2014 οι άνεργοι νέοι αλλά και οι νέοι που δεν είχαν τύχει καμία εκπαίδευση αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες και ο ρυθμός του ανήρχεται σε 6,5 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε φτάσει στα 7 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν ε, να ενθαρρύνουμε αυτούς τους νέους που έχουν χρόνο στη διάθεσή τους αλλά που δεν θέλουν να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη κατάρτιση όπως για παράδειγμα η μαθητεία. Πώς θα μπορούσαμε να τους ενθαρρύνουμε αυτούς τους νέους. Τι έχετε σκοπό να προτείνετε στον πρόεδρο Γιούνκερ για να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων λαθών. Θα πρέπει να υπάρξουν κοινωνικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα δίνουν προοπτικές και ελπίδες στους νέους. Θα πρέπει συνεπώς να επενδύσουμε στους νέους, όχι στις επιχειρήσεις, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Όχι, um, musím říct, že mm, přesně naplňujete το co si představuji, že by na úrovni Evropské komise... πάρα πολύ η παρέμβασή σας, κύριε Επίτροπε. Γιατί πραγματικά αυτό ήθελα να ακούσω να λέει η Επίτροπος. Ήθελα να ενημερωθώ για αυτό που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή για να διευκολύνει την μετάβαση από την εκπαίδευση στις ε, θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο γραμματικάκι. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές είναι θεωρητικές. Η κοινή ίση πρόσβαση είναι θεωρίες, αλλά οι οικονομικές αρχές θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν, αυτές που βρίσκονται στη βάση όλων αυτών. Ως επίτροπος Φαντάζομαι ότι θέλετε να επιτύχετε τους στόχους που προβλέπετε για το 2020, όπως τη μείωση των ε, μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Η Τσεχία πολλές φορές επικρίθηκε για το σχολικό δικό της σύστημα, ιδιαίτερα σε ό,τι τα παιδιά Ρομ. Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Επιτροπή θα μπορούσε να συμβάλλει στη λύση αυτού του προβλήματος. Η Τσεχία καταβάλει πολλές προσπάθειες για την ένταξη των παιδιών των Ρώμων η Τσεχία έχει το χαμηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα, γιατί τα παιδιά των Ρώμ βρίσκονται απομονωμένα, γιατί επικεντρώνονται με ένα δυσανάλογο τρόπο σε ορισμένα σχολεία. Αλλά ο μέσος όρος είναι πολύ καλός. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν ε, η, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Τσεχία κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την σαφήνεια των επιλογών της καταρχάς, για το γεγονός ότι υπογράμμισε ότι το βασικό μέλημα είναι η απασχόληση των νέων και μετά η ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι τα δύο αυτά σημεία κινούνται παράλληλα, αλλά θα πρέπει να γίνει μια επιλογή στον κοινωνικό τομέα. Κάτι απόλυτα σωστό. Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε κάτι και πιστεύω ότι θα να κάτι, κάτι εδώ η Επιτροπή. Ή στην Ευρώπη εδώ και καιρό υπάρχει πρόβλημα επενδύσεων. Αναφέρομαι στις ιδιωτικές επενδύσεις ιδιώτες τείνουν επενδύουν αλλού, γιατί υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι, λιγότερα προβλήματα ασφάλειας, ε, υπάρχουν προαπαιτούμενα που δεν υπάρχουν ε, αλλού. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να υπάρξει κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη όθηση στην επένδυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην Ευρώπη και όχι αλλού. Ξέρω ότι είναι μια δήλωση επιθεμάτων αρχής, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα και σε επίπεδο επικοινωνία. Είναι ένα από τα σημαντικά θέματα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την αξιολόγηση που κάνετε σχετικά με τον ρόλο της επαγγελματικής ε, κατάρτισης ε, και την ε, επαναφορά των παιδιών στα σχολεία. Αυτό όμω αυτή η ανάκτηση περνάει και μέσα από την αναγνώριση οικονομικού χαρακτήρα ε, που αφορά μια σειρά από εργασιακέ ε, δραστηριότητες στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που τίνουμε να υποτιμάμε. Το θέμα της εγκατάλειψης του σχολείου, το θέμα της διαβίου, παρακαλώ τελειώνετε. Τελειώνω, τελειώνω γιατί υπάρχει ένα ερώτημα που θέλω να κάνω. Εδώ και καιρό έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά υπάρχει ένα είδος αναντιστοιχίας ε, των ετοιμάτων που προέρχονται από την αγορά εργασίας για να προωθήσουν την ένταξη. Μία σειρά από επαγγέλματα που αφορούν το μέλλον και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε καν το περιεχόμενό τους και συμφωνώ μαζί σας, το ερώτημα που θέλω να κάνω, μήπως θα ήταν σκόπιμο αυτή τη στιγμή να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για μια καλή γενική κατάρτιση για να αποφευθεί η απόρριψη από την αγορά εργασίας όταν ακολουθούν οι διαδικασίες σαν και αυτές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γλέζος, ο συνάδελφος Χόλμερ και τελειώνουμε. Goedemorgen, mevrouw commissarin. Ως ε, αδαής ακροατής θαυμάζω την εισήγησή σας. Ως υπηρέτης 7 επιστημών και διδάκτορας 4 επιστημών από αυτές ερωτώ γιατί δεν ελαττώνεται η ανεργία έως τώρα, γιατί συνεχίζεται ακόμα η μετανάστευση. Και ηλικιακά ως σας δεν σας δίνω καμιά συμβουλή. Σας λέω μονάχα ένα παράδειγμα. Έχω συζητήσει με πάνω από 400 σχολεία στην πατρίδα μου. Σε κάποιο από αυτά τα σχολεία είπαν στο μαθητή όταν θα έρθει ο κύριος Γράζος να βγάλει το σκουλαρίκι σου δίσταζα γιατί το ήθελα να το φορώ και τελικά υποχρεώθηκα να το βγάλω και να σας ακούσω. Όταν σας άκουσα κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να το βγάλω. Άρχισα αλληλογραφία μαζί του και τελικά του είπα εάν το σκουλαρίκι το φοράς ως εναντίωση στο καθεστώς καλά κάνεις. Τον γονιό σου, των δασκάλων σου, παντού. Εάν το φοράς ως επίδειξη κάνεις κακό. Δεν σας συμβουλεύω, σας παρακαλώ μελετήστε αυτήν την άποψη. Ευχαριστώ. Collega Holbeni, prego. Holbeni, I don't know the Thanks a lot. That's right. Tisztelt biztos asszony, a kultúrát kicsit szét Ευχαριστώ πολύ. Αν κάνουμε μία ευρεία ερμηνεία του πολιτισμού, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται, περιορίζει εν μέρει αυτή την κινητικότητα. πολλοί νέοι μετακινούνται από τις νέες χώρες μέλη στις παλιές για να βρουν μια θέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι περιορισμένη, παρεμποδίζει την αναχώρηση από τις νέες χώρες μέλη και μιλάμε για τους εργαζόμενους στο υγειονομικό τομέα που μαζικά εγκαταλείπουν τις χώρες τους και προκαλούν μια αντί, ένα αντίστροφο dumping. Οι παλιές χώρες μέλη προσπαθούν να προσλάβουν εργαζόμενους από τις νέες χώρες μέλη στον υγειονομικό τομέα δίνοντας μισθούς που είναι υψηλότεροι από αυτούς που θα έπαιρναν στην παρατήρα τους και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο υγειονομικό σύστημα, στο σύστημα υγείας των νέων χωρών. Ελπίζω η Επιτροπή Γιούγκερ να μπορέσει να παρέμβει και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι έχει σκοπό να κάνει η Επιτροπή για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Μας είπατε ότι θα πρέπει να φύγετε αρκετά σύντομα. Σας είμαστε ευγνώμονες που παραμένετε λίγο περισσότερο πέρα από το πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ. Τα χαιρόμουν ιδιαίτερα να μπορέσω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση μαζί σας, αλλά με περιμένει ένας βουλευτής σε μια άλλη επιτροπή. Ενημερωτή Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στάζ, την πρακτική εξάσκηση στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τα διακρατικά στάζ, υπάρχει το σύστημα ΕΟΡΕΣ που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε. και μέσω του ΕΟΡΕΣ θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουν ε, οι ενδιαφερόμενοι να βλέπουν που, υπάρχει, που υπάρχουν ανάγκες. Θα πρέπει βεβαίως να είναι ορατές και οι θέσει τάζ έτσι ώστε να μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί το έουρες αν, αν ε, κάποιος αναζητάει μια θέση εργασίας στο εξωτερικό. Κύριε Νέκο, οι νέοι που δεν θέλουν να ακολουθήσουν μια ε, περίοδο κατάρτισης ή να βρουν μια θέση εργασίας. Δίχως άλλο, μπορούν να εργαστούν ως εθελοντές. Ενδεχομένως μερικοί από αυτούς δεν θέλουν ούτε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να εξυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Πολύ συχνά αυτό προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις γιατί θα πρέπει να διασπαλίσουμε ένα εξαίρετο σύστημα κοινωνικής προστασίας όταν μιλάμε όμως για εξυγχρονισμό, δεν θέλουμε να μειώσουμε τα δικαιώματα. Ο στόχος μας είναι να ορίσουμε το σύστημα έτσι ώστε να δημιουργεί ένα κίνητρο για τους πολίτες για να κάνουν κάτι. Θα πρέπει να έχουν μια όθηση, ένα κέντρισμα. Αυτό ισχύει και για αυτούς τους νέους. Δίχως άλλο θα υπάρχουν πάντοτε οι νέοι που δεν έχουν την διάθεση, που δεν έχουν τα προσόντα για να ενταχθούν σε αυτό το κύκλωμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με κοινωνικά κονδύλια. Αν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα απαραίτητα ε, τις δεξιότητες θα μπορούσαν να συμβάλλουν. Ας πούμε σκέφτομαι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν. Κύριε Τώρα, σχετικά με την Τσεχία και τους Ρωμά. Θέλω να σας πω ότι είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Ε, είμαστε λοιπόν ανοιχτοί στο θέμα. Βεβαίως και πρόκειται για μια ειδική ομάδα αυτή η ομάδα των Ρωμά και πολύ εύκολο ε, είναι να λέει κανείς κάτι όταν δεν τον αφορά. Αυτοί όμως που τους αφορούν γνωρίζουν ότι ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που δείξατε το θέμα αυτό. Βεβαίως και χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη και τις ε, επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο πλαίσιο επενδύσεων και με το πρόγραμμα Juncker θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε βελτιώσεις. Πάντως το πρόγραμμα επενδύσεων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όπως ξέρετε είναι πρικοδοτημένο με 350 δισεκατομμύρια. Εκείνο που επίσης θέλω να πω είναι ότι η πρόθεσή μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να άρουμε φραγμούς και να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη εσωτερική αγορά, κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Η ψηφιακή αγορά πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα. Πάντως αυτά είναι εκείνα που μας ενδιαφέρουν. Ορισμένες επιχειρήσεις ε, δεν είναι ακόμα έτοιμες ε, και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις παραδείγματος χάρη στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, ε, της κοινωνικής προστασίας. Εκεί πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις, να αφαιρέσουμε εμπόδια Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε πράγματι μια ισόρροπη λύση. Και κάτι άλλο που θέλω να πω ε, σχετικά με τη μετανάστευση. Γιατί δηλαδή εξακολουθούμε να έχουμε τόσους πολλούς μετανάστες. Α, ναι, το θυμήθηκα. Ε, αναφερθήκατε στους ε, τομείς της ε, υγείας ε, και μετα... αυτό σε σχέση με τη μετανάστευση. Βεβαίως ε, και όλοι έχουν το δικαίωμα της κινητικότητας, ε, της ελεύθερης μετακίνησης. Αυτό ε, είναι κατοχυρωμένο στις ιδρυτικές συνθήκες. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα της Ευρώπης ε, να πει στους ανθρώπους «Ξέρετε, θα μείνετε εκεί που γεννηθήκατε». Μα δεν είναι έτσι. Ε, βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και ε, μπορεί κανείς να διασχίσει τα σύνορα, αλλά θα πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικός με τα προβλήματα που υπάρχουν, τις ευαισθησίες που υφίστανται. Αυτές οι ευαισθησίες σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι πολύ πιο έντονες από ό,τι σε άλλα. Ε, εκείνο που παίζει επίσης ρόλο είναι να δούμε τι διαδραματίζεται στα κράτη-μέλη. Εγώ εκείνο που προσέχω πάρα πολύ είναι να εντοπίζω τις ευαισθησίες, να ξέρουμε που πρέπει να κινηθούμε, αλλά το να περιοριστεί η κινητικότητα νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Εγώ πρέπει να σας πω ότι μεγάλωσα με την κοινή αγορά και την ελεύθερη μετακίνηση και αυτό δεν θα το περιορίσουμε μόνο για εμπορεύματα και αγαθά. Αν θέλουμε να περιορίσουμε τους ανθρώπους, ε, τότε να περιορίσουμε και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που αυτά είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα δούμε πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα και κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να επιφέρουμε βελτιώσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά που είπατε ήταν πολύ σημαντικά και η ειλικρίνεια με την οποία μιλήσατε. Έτσι λοιπόν ας παραμείνουμε με το μήνυμα που προέκυψε από πολλούς συναδέλφους ότι η προτεραιότητα της απασχόλησης θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται και με το, από το θέμα των προσόντων. Ε, και της γενικότερης παιδείας γιατί αυτό είναι το μόνο εργαλείο για να έχουμε καινοτομία και ευθύη ανάπτυξη. Επίσης ε, στο θέμα των επενδύσεων Juncker όπως ακούσαμε γίνεται λόγος ε, γενικότερα για την παιδεία όμως δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα ο πολιτισμός. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και εύχομαι με τον τρόπο αυτό να έχουμε μια αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίγο αυτό που είπε και ο κύριος Γραμματικάκης, δηλαδή να δώσουμε νέα πρότυπα, μια νέα φιλοσοφία, ε, να μην μιλάμε έτσι γενικά και αφηρημένα για την ανάπτυξη, γιατί αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα υποκείμενα δεν υπάρχει και ανάπτυξη. Λοιπόν, συνάδελφοι, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λόγω του ότι τα απόγευμα στις 3 ώρα τα έχουμε ακρώσει. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική έκθεση ε, της συναδέλφου ε, Κριστίνα Λιμπάκα. Πρόκειται για τη συνέχεια που δόθηκε στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Θα θυμάστε ότι η τελευταία υπουργική συνδιάσκεψη ε, σχετικά με αυτά τα θέματα έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι το 2012. Και η επόμενη συνάντηση των υπουργών θα λάβει χώρα το Μάρτιο του 2015 στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Κατόπιν τούτου, αυτή η δουλειά που έχει κάνει η συνάδελφο, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η συνάδελφος, το λέω αυτό και υποκλίνομαι γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, με πολύ καλή συνεργασία, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας. Τώρα λοιπόν έχουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να εξεταστεί πριν από τη συνάντηση των Υπουργών. Να επενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Διορία για τις τροπολογίες. Όπως αναφέρθηκε ήδη μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ε, και μην ξεχνάτε την 24η Μαρτίου που είπα για τη συνεδρίαση των Υπουργών. Πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν γινόταν αλλιώ. Ε, δεν θα προλαβαίναμε να καταθέσουμε την έκθεσή μας. Συνάδελφε, κυρία Λιμπάτσκα, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω όπως Εξάλλου και στο κείμενό μου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και ευχαριστώ πραγματικά όλους τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτήν την διαδικασία της Μπολόνια και έχουν συνεισφέρει με την εμπειρία τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους σπουδαστές, τους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ όλα τα κράτη-μέλη που υπέβαλαν σχόλια και παρατηρήσεις. Ήμουν ε, δυστυχώς περιορισμένη στην ε, πρότασή μου όσον αφορά τον αριθμό των λέξεων, το μέγεθος αυτής της πρότασης. Εγώ η ίδια υπέβαλα κατόπιν 20 τροπολογίες Πολλές από αυτές βεβαίως είναι κοινέ τροπολογίες γιατί λαμβάνουν υπόψη και απόψεις άλλων. Αν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες ή να ε, σχολιάσετε κάποια από αυτές, φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μου. Φυσικά και ο τομέας αυτός χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις και προσθήκες. Οι 15, τα τελευταία 15 χρόνια στα οποία λειτουργήσε η διαδικασία της Μπολόνια είδαμε βελτίωση της κινητικότητας, νέες ε, ακαδημαϊκές δομές και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα τομείς που θα πρέπει να ενισχυθούν. Η διαδικασία της Μπολόνια αντιμετωπίζει σήμερα και νέες ε, προκλήσεις καθότι η πραγματικότητα διαρκώς εξελίσσεται και αλλάζει. Τι είναι καινούριο καταρχήν σε αυτή τη διαδικασία. Όλα τα κρατημέλη αποφάσισαν να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος, μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να καταργήσουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Χρειάζεται λοιπόν να εντοπίσουμε τις προσπάθειές μας στην διδασκαλία. Αυτό έχει ήδη γίνει, αλλά χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια. Χρειάζεται, αν θέλετε, διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης και η διδασκαλία, η έννοια της διδασκαλίας, αν θέλετε, πρέπει να βασίζεται στην ερώτηση τι γνώσεις χρειάζονται οι μαθητές και οι φοιτητές σήμερα. Κάτι άλλο που θα πρέπει σαφώς να προσέξουμε, πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται σήμερα, είναι το θέμα της ε, αναγνώρισης ε, ξένων δεξιοτήτων και πτυχίων, ο τρόπος που αξιολογείται και λαμβάνεται υπόψη η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό. Η άτυπη αλλά και επίσημη εκπαίδευση πώς λαμβάνεται υπόψη. Το θέμα των credits, της πιστοποίησης, αλλά και βεβαίως η διαβίου μάθηση. Ένας άλλος τομέας που θα πρέπει σαφώς να εξεταστεί είναι το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν αποφάσεις για την αναγνώριση, παραδείγματος χάρη, των πτυχίων τους μέσω τρίτων ανεξάρτητων οργανισμών και φορέων. Βλέπουμε επίσης τα ανώτατα ιδρύματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν παίζουν πολλές φορές το ρόλο τους αναγνώρισης και πιστοποίησης των πτυχίων και των δεξιοτήτων. Το θέμα επίσης της πρακτικής άσκησης, των στάζ στην Ευρώπη. Φυσικά και αυτό είναι κάτι που το συζητούμε σε πολλές λεπτομέρειες και εις βάθος. Πολλές χώρες έχουν εντοπίσει ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι κάτι που σαφώς ε, ανταποκρίνεται σε ανάγκες της ε, σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η αναγνώριση μίας περίοδου σπουδών στο εξωτερικό ή στην ίδια τη χώρα, η ενσωμάτωση του ECTS, το θέμα της ε, πρώτης περίοδου κατάρτισης αλλά και των μεταγενέστερων, η διαδικασία της Μπολόνιας καθώς και τα κοινωνικά εμπόδια που συνεχίζουν να υπάρχουν. Η διεθνής κινητικότητα για κάποιες ε, κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κοινωνικές ομάδες που δεν εκπροσωπούνται όπως θα έπρεπε στη διαδικασία της Μπολόνια και στην κινητικότητα. Αυτές τις κοινωνικές ομάδες πρέπει να τις ενισχύσουμε. Πρέπει επίσης να υπάρξουν και διεθνές ε, μελέτες αλλά και διατομεακές μελέτες και έρευνες όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της ε, Μπολόνια. Το θέμα επίσης της απασχολησιμότητας, του επίπεδου της ε, απασχόλησης. Η εκπαίδευση βεβαίως καταρχήν είναι η μετάδοση γνώσεων στους φοιτητές και στους μαθητές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την συνολική προσέγγιση που έχουμε προς τους μαθητές και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της έρευνας, της μετάδοσης γνώσεων, της γενικότερης ανάπτυξης των φοιτητών και μαθητών και βεβαίως των σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας, επιχειρήσεων. Η διαδικασία της Μπολόνιας πώς θα πρέπει να ενισχύσει και τον... την όλη πρωτοβουλία έρασμους και βεβαίως τους ε, στόχους του Horizon 2020. Είναι αυτονόητο ότι εμείς θα πρέπει να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να δούμε και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων, εντοπίζοντας βεβαίως νέους τρόπους χρηματοδότησης και νέες πηγές χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους αδέλφους που το ζήτησαν Σβέρ, Μάουρα και Μαραγκάλ. Σε αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριος Σβέρ, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πάρα πολύ καλή της έκθεση, την κυρία Κριστίνα Λιμπάτσκα. Και είμαι πεπισμένος ότι η αγαστή συνεργασία με όλους τους ε, σκιώδης θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλή τελική έκθεση σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια. Όσον αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια, ακούσαμε πάρα πολλές ε, και καλές εκθέσεις. Ας πούμε, ο κύριος Μπελιγκουέρ ε, προτίμασε ε, πάρα πολύ καλή έκθεση πριν από τρία χρόνια. Εν τω μεταξύ όμως, η έκθεση αυτή πραγματικά είναι ακόμα καλύτερη και ιδιαίτερα επίκαιρη. Όσον αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια, αυτή αφορά 47 ε, χώρες, ε, το Συμβουλίο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχολικές ε, ενώσεις, κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή μία σειρά διαφορετικούς εμπλεκόμενους που συμμετέχουν σε αυτή την τόσο σημαντική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 17 χρόνια. Τότε είχαμε κάποιους από τους οραματιστές οι οποίοι ε, δρομολόγησαν τη διαδικασία. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για πάνω από μία δεκαετία ε, κατορθώσαμε πάρα πολλά σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Περάσαμε μέσα από αυτούς τους ε, τρεις κύκλους αλλά εισαγάγαμε και μία σειρά μηχανισμών που επέτρεψαν στα ευρωπαϊκά, να υπάρξουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ένας ευρωπαϊκός ε, χώρος. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα χώρο που μπορούν να γίνουν συγκρίσεις. Εξάλλου υπάρχει και το ε, Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Ε, υπάρχει έλεγχος, ε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων, το οποίο βέβαια ακόμα εκκρεμεί ως προς την ε, θέσπισή του σε εθνικό επίπεδο. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι τα προγράμματα των πανεπιστημίων, προγράμματα εντασκαλής. Αυτά είναι πολύ πιο εύκολο να συγκριθούν. Και σε επίπεδο περιεχομένου έχουμε επιτύχει πάρα πολλά σε τεχνικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά στην αναγνώριση των διπλωμάτων και των άτυπων δεξιοτήτων. Ξέρετε, ο ακαδημαϊκός χώρος ε, θα πρέπει εδώ να κάνει πολλά περισσότερα. Κυρίως ε, στον ε, τομέα των λυκείων και των πανεπιστημίων. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην εισαγωγή των πολυεθνικών στο ρόλο που παίζουν στις διάφορες χώρες ε, παραδείγματος χάνη της McDonald's, ε, της Siemens, ε, της Volkswagen υπάρχουν συστήματα που εφαρμόζουν πολυεθνικές που δεν είναι όμως αναγνωρισμένα. Όσον αφορά τώρα τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας της Μπολόνια και το σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο. Πλέον υπάρχουν ε, δεξιότητες ε, οι οποίες όμως δεν ε, επικρατούν σωστά σε κοινωνικό επίπεδο. Έχουμε πάρα πολλούς άνεργους. Έχουμε ανεργούς αλλά απ' την άλλη έχουμε και θέσεις που δεν καλύπτονται. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάπου υπάρχει μια αναντιστοιχία θέσεων απασχόλησης με δεξιότητες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στην επιστήμη, στα μαθηματικά, στη μηχανολογία. Όλα αυτά ε, θα πρέπει να καταστούν ε, πιο ελκυστικά για τους νέους, διότι ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται αυτούς τους εμπειρογνώμονες, χρειάζεται συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Και μερικές φορές πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια απλά είναι πολύ εξαρτώμενα από το κράτος. Και αυτή είναι η μορφή ε, πανεπιστημίων που ε, βρίσκονται σε ύφεση. Τώρα ε, εμφανίζονται σιγά σιγά τα ανοιχτά πανεπιστήμια που μπορούν να πουλήσουν την τεχνογνωσία στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτά τα ανοιχτά πανεπιστήμια είναι πολύ πιο στενά συνδεμένα με τις παγκόσμιες τάσεις. Τελειώνω, τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να πω ότι η επόμενη γενιά των πανεπιστημίων ε, θα είναι ανεξάρτητη, γιατί η επόμενη γενιά θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς την επιρροή της κρατικής γραφειοκρατίας. Η έκθεση της κυρίας Λιμπάτσκα νομίζω ε, θα φέρει προς τη θέμενη αξία και θα έχει θετικές επιπτώσεις στην περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας της Μπολόνια. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε. Ε, επόμενος ερωτών ή ερωτώσα, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Κυρία Πρόεδρε, ε, θα είμαι σύντομος, λέει ο κύριος Μάουρα. Καταρχήν ευχαριστώ την κυρία Λιμπάτσκα και άλλους και ηγητές για αυτή την έκθεση ε, σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά ε, και η προετοιμασία ήταν πολύ καλή στην Επιτροπή Πολιτισμού προσπαθούμε να προβούμε σε απολογισμό και να δούμε γενικά τι διαδραματίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς έχουν αλλάξει τα ε, συστήματα της ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, εκπροσωπούμε τους πολίτες, γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η παιδεία είναι το σημαντικότερο εργαλείο για να μπορεί κανείς να εξελιχθεί περαιτέρω επαγγελματικά και κοινωνικά. τα πανεπιστήμια έχουν αλλάξει στην Ευρώπη με μεταρρυθμίσεις και αυτό είναι πολύ καλό. Έχουν υπάρξει αλλαγές και για το διδακτικό προσωπικό και για τους ε, φοιτητές. Τώρα πια υπάρχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα, υπάρχει συμπληρωματικότητα. Αυτό προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές που είναι και πιο κινητικοί διότι αναγνωρίζουν τα πτυχία τους. Όμως πρέπει να καταβάλουμε και άλλες προσπάθειες να μεριμνήσουμε να επιτευχθούν οι εξή στόχοι. Πρώτον, ε, ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους. Δεύτερον, απασχολησιμότητα για όλους να τη διασφαλίσουμε αυτή κατόπιν, ε, να υπάρχει καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Εμείς έχουμε συμβάλει σε αυτή την έκθεση με την κατάθεση τροπολογιών με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, προαγωγή της αναγνώρισης πτυχίων και πέρα από τα σύνορα, διασυνοριακά δηλαδή. Δεύτερον, διατήρηση ποιοτικών προδιαγραφών ε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τρίτον, εγγυήσεις διαφάνειας, αυτό μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο παιδείας. Όσον αφορά τώρα στη στρατηγική που εφαρμόζουν τα πανεπιστήμια, αυτή είναι σημαντική για την κοινωνική ενσωμάτωση και για την απασχόληση. Και τελειώνοντας, το 1990 είχαμε μια κοινή δήλωση για τη διαδικασία της Μπολόνια και αυτή ήταν και η έκρηξη που δημιούργησε τον Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Χώρο. Η επέκταση αυτού του χώρου είναι ευκαιρία και καθήκον για μας για να μπορέσουμε να προάγουμε τις αξίες τις οποίες μεριζόμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Πολύ ωραία, συνάδελφος Μαραγκάλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, δεν προβλέπονται τα καταλανικά για τη διερμηνία και γι' αυτό ε, θα μιλήσω ισπανικά. Τι να κάνω θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα στην Ισπανία έχουμε μία διαμαρτυρία. Αφορά στις τελευταίες αποφάσεις που ελήφθησαν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διαδικασία της Μπολόνια. Εκεί γίνεται λόγος για δηλαδή, τα διάφορα πτυχία, το bachelor, το master. Σε πολιτικό επίπεδο, όσον αφορά αυτή τη διαμαρτυρία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η διαδικασία της Μπολόνια δεν έχει εμπνεύσει σεβασμό, τουλάχιστον όχι σε εμά στην Ισπανία. Και γι' αυτό δεν υπήρξαν και πολλές ε, θετικές επιπτώσεις στην Ισπανία από αυτή τη διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη συνέχεια αλλά να υπάρξουν και κάποιες ε, βελτιώσεις. Και νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος της συνάντησης που θα λάβει η χώρα το Μάιο. Όσον αφορά την οργάνωση και το περιεχόμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ε, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ποιοτικό πλαίσιο για την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε ανισορροπίες που υπάρχουν στον χώρο των πανεπιστημίων. Επίσης, να πλησιάσουμε το στόχο μας. Πριν από 15 χρόνια είπαμε ότι θέλουμε έναν ευρωπαϊκό ε, χώρο ε, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ποιότητα, ελευθερία, διασύνδεση με την κοινωνία. Νομίζω θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό το ότι πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι κατά πόσον τα πετύχαμε όλα αυτά ε, και βέβαια να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα ως εκ τούτου. Να δούμε τι έχουμε πετύχει και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Λιμπάτσκα, την εισηγήτρια, για τη δουλειά της, για το διάλογο που είχε όχι μόνο με την πολιτική ομάδα αλλά γενικότερα με τον ακαδημαϊκό κόσμο και με τους φοιτητές. Εμείς ε, έχουμε καταθέσει πολλές τροπολογίες, τις επεξεργαστήκαμε από κοινού. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ε, προσθήκες. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές, καθοριστικές για μένα, ε, πάντα σε σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνια. Πρώτον, αυτό που ενδιαφέρει είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, όχι η διοίκηση, να γίνεται σεβαστό το Πανεπιστήμιο. Κατόπιν, χρειαζόμαστε ένα πραγματικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Τρίτον, πρέπει να υπάρχουν βασικοί δείκτες και όλοι να τους ενστερνιστούν αυτούς για να υπάρχουν και διορθώσεις και βελτιώσεις στη διαδικασία. Τέταρτον, θα πρέπει να περνάμε από μια καθαρά τυπική σε μια ουσιαστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ε, χρειαζόμαστε ε, ε, μεγαλύτερη λογοδοσία Τελευταία μου παρατήρηση, λέει ο μιλητής, η οικονομική κρίση οδήγησε σε πολλά προβλήματα όσον αφορά στην εφαρμογή της διαδικασίας. Γι' αυτό να υπάρχουν ε, κριτήρια σύγκλησης, ε, κυρίως ε, αν δεν θέλουμε να υπάρχουν διαφορές. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εγώ θέλω να παρακαλέσω του αντέλφου να λαμβάνουν υπόψη στο χρόνο που διατηρείτε. Κύριε Γλέζο, εσείς έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, η παιδεία είναι δικαίωμα ιερό και πρέπει να παρέχεται σε κάθε πολίτη πλούσιο ή φτωχό είτε ανήκει σε θρησκευτική είτε φιλετική μειονότητα. Αυτό πρέπει να είναι το, ο κύριος στόχος μας και έτσι πρέπει να διασφαλίζεται από την πλευρά μας, ο ένας τομέας. Ο δεύτερος τομέας είναι ότι πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση ο οποιοσδήποτε φοιτητής στο κύκλο των, των σπουδών του. Εδώ υπάρχει ένας περιορισμός που αποσκοπεί στην ικανοποίηση μόνο της αγοράς και όχι του ιερού δικαιώματο της παιδείας και αυτό που λέμε κατά κόρον και δεν γίνεται στην πράξη διαβίου μάθησης. Στην Ελλάδα τώρα που ήρθε μια κυβέρνηση πριν από ένα μήνα όπου ο λαός παίρνει την τύχη του στα χέρια του θα εφαρμόσει μια πραγματική παιδεία και θα ήθελαμε και τη βοήθεια σας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Grazie collega Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Απλά ε, να πω το εξής. Ε, υπάρχει ουσιαστικός βαθμός συνεργασίας και προσαρμογής και αυτό συνεχίστηκε με την έκθεση. Ε, πολλοί συνυπέγραψαν και αυτό δείχνει ότι πολλοί συμφωνούν. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια γι' αυτό. Βεβαίως... Ε, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν όλα αυτά, θα ήταν και παράλογο. Κάποιος από την Κομισιόν μίλησε για κάτι ιδιαίτερα θαραλέο, μου είπε κάτι πολύ θαραλέο και ενδιαφέρον που είναι από λίγες ημέρες. Δηλαδή, ε, μια έκθεση επί της οποίας συμφωνούν όλοι, η υπερβολική συνένεση, ε, είναι και προβληματική, δεν είναι καλό πράγμα. Εγώ νομίζω ότι στην έκθεση αυτή Έχουμε προχωρήσει πολύ. Οι αντιφάσεις ανάμεσα ας πούμε, στο, στην αυτονομία των πανεπιστημίων και την ε, κρατική ε, ρύθμιση υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να επιληθούν και κάπως επιλύονται νομίζω στην έκθεση αυτή. Κάτι που δεν έχει γίνει ε, σεβαστό είναι η επόμενη φάση της διαδικασίας της Μπολόνια. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αποδίδει σημασία όχι τόσο στο περισσότερο, όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα. Η αυτονομία είναι λέξη κλειδί, πολύ σωστά. Το πρόγραμμα Erasmus Plus ε, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο ακόμα και οι ευρωσκεπτικιστές μεταξύ μόν μπορούν να το στηρίξουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Ε, και τέλος κάποια σχόλια που έκανε η κυρία Λεμπάτσο και άλλοι για το πρόγραμμα Horizon 2020. Ε, πολύ σημαντικό. Ε, εδώ θα έρθουν ακόμα πολλά. Πολλοί ανησυχούν για το ότι υπάρχουν κάποιες κερδοσκοπικές επενδύσεις που δεν γίνονται βέβαια από το κράτος. Τέλο πάντων, θα υπάρχουν ε, πάρα πολλά ακόμα στο μέλλον. Επειδή όμω θέλω να σεβαστώ το χρόνο που μου δώσετε, κυρία Πρόεδρε, τα δύο λεπτά και δεν θέλω να τον υπορβώ, εγώ ε, σταματάω και ελπίζω το παράδειγμά μου να το ακολουθήσουν και άλλοι. Thank Σύντομη θα είμαι. ευχαριστώ. Θα ήθελα Να σας ε, ευχαριστήσω, καταρχήν ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Τα σημεία 12 και 13 είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την ε, Επιτροπή και θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ, και το λέω αυτό στην εισηγήτρια, με κάποιες τροπολογίες. Θεωρώ πραγματικά ότι αυτή η διαδικασία της Μπολόνιας καθώς και η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν είναι κάτι που θα πρέπει να μας κάνει πιο προσεκτικούς όσον αφορά την ε, υλοποίηση των ε, κανόνων, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την αναγνώριση των ε, διπλωμάτων και των πτυχίων. Παραδείγματο χάρη στην Ουκρανία υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να διδάξουν μέχρι να πάρουν την τοπική πιστοποίηση, από όπου και αν προέρχονται. Εγώ πήρα το διδακτορικό μου στην Βουδαπέστη και αναγκάστηκα να επαναλάβω όλη μου την εργασία στο Κίεβο, αλλιώς δεν μπορούσα να διδάξω. Οι αρχές στην Ουκρανία ήθελαν κάθε φορά να εξετάσουν με δικά τους κριτήρια και με δικό τους τρόπο την διάκριση, το δίπλωμα, το πτυχίο που κάποιος είχε πάρει κάπου αλλού. Νομίζω ότι όμως σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος συμμετέχει στη διαδικασία της Μπολόνιας, θα πρέπει να δέχεται τους κοινού μας κανόνες και να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Όπως υποστηρίζει η έκθεση, η διαδικασία της Μπολόνια επιτυχάνει τους στόχους της για την αναγνώριση των τυπικών προσόντων, θα πρέπει να γίνει και κάτι περισσότερο. Θα πρέπει να βελτιωθούν τα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να μετρηθεί η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της απασχολησιμότητας και της απασχόλησης. Ο ρόλος των εργοδοτών θα μπορούσε να διεκρινιστεί περαιτέρω και κάτι άλλο, τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δεν θα ηγηθούν ποτέ της διαδικασίας της Μπολόνια αυτό είναι ευθύνη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ασκήσουν πιέσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια βελτίωση διαδικασία στην Πολόνια. Δεν θα περιμένω τα πανεπιστήμια να είναι εκείνα που θα παρέμβουν. Δίχως άλλο εμπλέκονται στην διαδικασία. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να στραφώ προς την εισηγήτρια και να της πω ότι πραγματικά την συγχαίρω και θα ήθελα να εντοπίσω τις παρατηρήσεις μου στο θέμα των διδασκόντων γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ να μιλήσουμε για την ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας. Νομίζω ότι η διαδικασία της Μπολόνιας θα πρέπει σαφώς να ενισχύσει αυτή την ελευθερία και να εντοπίσει ιδιαίτερη προσπάθεια στην έρευνα που λαμβάνει η χώρα στο εσωτερικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε αντιπαράθεση με την έρευνα που χρηματοδοτείται και γίνεται από τις επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να διατεθούν λοιπόν κονδύλια και για να διασφαλίσουμε αυτήν την έρευνα. Η ελευθερία των καθηγητών της διδασκαλίας. Εδώ δεν αναφέρομαι μόνο λοιπόν στην ελευθερία του ίδιου του καθηγητή ή του ε, διδάσκοντα, αλλά στην ελευθερία που πρέπει να έχουν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έτσι ώστε να επιλέξουν τους τομείς αυτούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Να υπάρχει δηλαδή μία ε, αν θέλετε ελευθερία που να επιτρέπει την συμμετοχική διδασκαλία. Κάτι που βλέπουμε σήμερα να μην ε, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας. Πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε και σε αυτό να το υπογραμμίσουμε γιατί είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και δεν θα πρέπει μόνο να στοχεύουμε τις προσπάθειές μας σε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνολογικά θέματα, αλλά και σε αυτά που σίγουρα θα πρέπει να εμπνέουν την κοινωνία μας, που είναι η πραγματική συνεισφορά της ακαδημαϊκής κοινότητας των καθηγητών για μια κοινωνία που θέλουμε να γίνει καλύτερη και η έρευνα σίγουρα θα πρέπει εδώ να ενισχυθεί στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια με την έννοια ότι σήμερα κινδυνεύουμε να περιορίσουμε ιδιαίτερα αυτούς τους τομείς που δεν είναι επιστημονικοί, που δεν είναι τεχνολογικοί, κάτι που μπορεί να διακινδυνεύσει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ο συνάδελφος Μόργανο. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ και εγώ για τα όσα έκανε άνθρωση Κατερίνα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία. Η στρατηγική σημασία της διαδικασίας στην Πολόνια επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, τις ε, αναφορές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που έγιναν την τελευταία 15 ετία καθώς και τις νέες προκλήσεις. Έχουμε προβλήματα οικονομικής κρίσης, δημογραφικών αλλαγών, εσωτερικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τρομοκρατία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, αγνοήσουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα της κατάρτισης. Είναι σαφές και θα πρέπει να το τονίσουμε για μία ακόμα φορά, αλλά προκύπτει και από τα όσα υπόθηκαν, υπάρχει μια πολιτική πτυχή στην εμπλοκή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων καθώς και των άλλων παικτών σε μια προσπάθεια να γίνουν τα απαραίτητα βήματα. Είναι ανώφελο να μιλάμε διαφορετικά για ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της αξιολόγησης των συστημάτων κατάρτισης Δηλαδή θα πρέπει να καταβληθεί μια προσπάθεια να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότερα δείγμα, ε, ε, δίκτυα μεσίτοβροβαρικά για να γίνουν περαιτέρω βήματα. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει κάτι να μας πει. Θα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την κυρία Λιμπάτσκα για την έκθεση ε, για το σχέδιο έκθεσης που εστιάζεται στα βασικά θέματα που έχουν σχέση με την προετοιμασία της συνάντησης των Υπουργών τονίζεται το θέμα της εφαρμογής, όπως είπε ένας συνάδελφος, το πώς θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όχι να κάνουμε περισσότερα. Νομίζω ότι εκεί η κατάσταση διαφέρει μεταξύ μας. Βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να πάψουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές που ανέκυψαν μετά τη διαδικασία της Μπολόνια, ιδιαίτερα την επίπτωση της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη της αύξησης ε, της απασχολησιμότητας των ε, πτυχίουκων καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο νέο είδος ε, φοιτητών, τους οποίους αφορά η ανώτατη εκπαίδευση. Θα πρέπει δηλαδή να στηρίξουμε τα πανεπιστήμια στην προσπάθεια ανάπτυξης ψηφιακών μέσων μάθησης και ε, Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να συνδυαστεί η έρευνα με τη διδασκαλία, με τη μάθηση για τους ε, μαθητές. Και αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τις ανάγκες, τις αμυγείς ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε ό,τι με αφορά θα φροντίσω τα μηνύματα αυτά από το Κοινοβούλιο να γίνουν απόλυτα κατανοητά από τους εταίρους στην διαδικασία της Μπολόνια κατά την προετοιμασία για τη συνδιάσκεψη του Γερεβάνα. Και ελπίζω να υπάρξει γενικότερη συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Τάισεν. Η κυρία Λιμπάτσκα. Παρακαλώ. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy także dzisiaj. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι ακόμα και σήμερα σχολίασαν την έκθεσή μου με τις παρατηρήσεις αυτές. Έχω την εντύπωση ότι η συνεργασία μας ήταν πολύ επικοδομητική και ότι μπορεί κανείς να πει σήμερα ότι πρόκειται για μια κοινή έκθεση. Θα επικεντρώσω τα σχόλιά μου σε δύο μόνο σημεία, γιατί με τα υπόλοιπα συμφωνώ. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχει το πρόβλημα της χρηματοδότησης, όπως έλεγε ο συνάδελφος Κώσταρ. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης, γιατί όταν υιοθετήθηκε η διαδικασία της Μπολόνια είχαν ε, δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να δαπανίσουν το 3% του ΑΕΠ τους για το τομέα της εκπαίδευσης. Βεβαίως ε, αυτό δεν έγινε ποτέ και τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για την παιδεία είναι ανεπαρκή. Έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες ε, όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές δεξιότητες, την επιστημονική πτυχή της ε, παιδείας. Και εγώ συμφωνώ ότι πολλές φορές ε, εγκαταλείπουμε λίγο τις υπόλοιπες επιστήμες τις ανθρωπιστικές επιστήμες παραδείγματος χάρη, κάτι που εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μάλιστα πέρσι είχα κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την Πολωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι η γενικότερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ε, νέων μας είναι κάτι που θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Το θέμα τώρα της απασχολησιμότητας. Ναι, η συνεισφορά των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι καθοριστική, αλλά φυσικά οι θέσει απασχόλησης δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις, από την οικονομία και όχι από την εκπαίδευση τελικά. Ευχαριστώ αγαπητή Κριστίνα. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών αύριο στις 12 και στις 24 θα γίνει ψηφοφορία. Περνάμε τώρα σε μια άλλη γνωμοδότηση Νομοδότηση για την ε, έκθεση της Επιτροπής Γιούρη η γυρία Αντινόλφη τη συνέταξε και αφορά την αρμόζη ορισμένων πτυχών του δικαιώματο του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία τη πληροφορία. Η Επιτροπή Γιούρη θα ψηφίσει 16 Απριλίου. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμά μα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου. Όπως γνωρίζετε, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι αύριο στις 12. Συνάδελφος Ενόρτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι είμαστε υπέρ της ενιαίας ψηφιακής αγοράς η οποία αφορά 10 βασικά σημεία του προγράμματος Juncker. Είμαστε υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών και θεωρού, είμαστε υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει πρόθεση βασικών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία έκφρασης, σκέψης και γενικά στα όσα προβλέπονται από την Χάρτα των Βασικών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία είναι παροχημένη πλέον, δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η Επιτροπή η οποία εντοπίζει την ε, εντόπισε την προβληματική στο σάμιτ που έγινε στη, στη Λισαβόνα το Σεπτέμβριο του 2012. Με την ευκαιρία εκείνη, ο Κρός, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για την ψηφιακή ατζέντα, ζήτησε Αναφέρθηκε στο ρόλο που θα μπορούσαν να αναπέξουν τα, συγγενικά, δικαιώματα δημιουργού ή τα πνευματικά δικαιώματα. Η οδηγία InfoSoc είναι το τελευταίο εργαλείο που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στην Ηνωμένη Ευρώπη. Αλλά βασίστηκε σε όσα είχαν αποφασιστεί το 1998, ε, όταν ο Ζούκεμπεργκ που ανακάλυψε το ε, Facebook ήταν 14 ετών. Οι περισσότεροι ακούγαν μουσική στο, ε, από το ραδιόφωνο. Η ίδια, το ίδιο γεωγραφικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε ριζικά. Τώρα έχουμε να κάνουμε 28 ξεχωριστές χώρες. Πώς θα μπορούσαμε να περιμένουμε ξένες επενδύσεις, αν έχουμε να κάνουμε με 28 διαφορετικές νομοθεσίες, πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τους Αμερικανούς. Η ανάγκη εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα αναφέρεται ως στόχος στο πρώτο εκτιμώντας της ίδιας οδηγίας, σε ένα σχόλιο το οποίο λέει η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία ενός συστήματος που εγγυάται την απουσία εκτροπών του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η εναρμόνιση των νομοθεσιών των χωρών μελών σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Ορισμένα ερευνητικά κέντρα όπως το αυτό του Άμστερνταμ ε, παρομοίασαν την ανάπτυξη αυτού του τομέα που ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα με τα κλαδιά ενό δέντρου που θα πρέπει να κλαδεύονται. Η ίδια η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή μιλώντας για την βιομηχανία της μουσικής αναφέρει σαφώς ότι μέχρι σήμερα υπάρχει ένα σημαντικός ρυθμός αμφισημιών που δεν ε, ε, λαμβάνονται υπόψη στην οδηγία InfoShop και στις άλλες οδηγίες που ασχολούνται με το θέμα του copyright. Συνεπώς, στο φως όσων είπα μέχρι τώρα, καθίσταται ξεκάθαρη η ανάγκη να τροποποιηθεί η οδηγία InfoSoc για να προσαρμοστούν οι, οι δημιουργοί στις μικρές και μεγάλες χώρες, έτσι ώστε να επιτευθεί η κοινή ψηφιακή αγορά, η οποία προσεγγίζει τις ανάγκες των καταναλωτών. Το κίνημα των πέντε αστέρων κινείται και στηρίζει τους αδύνατους. Το θέμα της, των δημοτικών δικαιωμάτων μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Η ψυχολογική πίεση που οι εκπρόσωποι ιδιωτικών συμφερόντων άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή προβάλλοντας ε, μελέτες δεν αφήνει περιθώριο σε αυτό που είναι ο βασικός μας στόχος ως εκπροσώπου των πολιτών. Αυτό διακυβεύει την αυτονομία των επιλογών μας και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή για να υπάρξει η προστασία του κοινού αγαθού και την προστασία των πιο αδυνάτων που σε αυτή την περίπτωση είναι ε, ε, πολύ δημιουργή και βεβαίως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτές είναι αρχές που με οδήγησαν στο να συντάξω αυτή την γνωμοδότηση. Θα ήθελα τώρα, εν συντομία, να αναφερθώ στα διάφορα σημεία. Σημείο 1. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γίνει ένας ορισμός του δημόσιου χώρου και να υπάρξουν εξαφεί κανόνε για τα, δικαιώματα του δημιουργού. Θα πρέπει να συνοδεύεται αυτό από την υποχρέωση μη νομοθεσία. ε, όταν υπάρχει εναρμόνιση. Η έλλειψη κοινών κανόνων που αφορούν τα δικαιώματα του δημιουργού επιτρέπουν στις χώρε μέλη να παρεκκλίνουν από τους κανόνες που αφορούν τη διάρκεια των δικαιωμάτων του δημιουργού. Ε, δημιουργώντας προβλήματα για το δημόσιο χώρο και περιορίζοντας την κυκλοφορία της γνώσης σε κοινωνικό επίπεδο. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα αφορά το μικρό πρίγκιπα. Όταν μιλάω για δικαιώματα δημιουργού αναφέρομαι και σε συγγενικά δικαιώματα, το δικαίωμα των εκτελεστών, τα δικαιωματογραφικά, δισκογραφικά δικαιώματα. Απλά και μόνο για να αναφέρω μερικά. Σημείο 2 της γνωμοδότησης. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί το άρθρο 2 και 3 της οδηγίας για να διευκρινιστεί το θέμα του δικαιώματο αναπαραγωγή. Στο φω τη πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου, λαμβάνοντα υπόψη τι τεχνολογικέ Εξελίξει σε ψηφιακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Δερκή προσανατολισμό του δικαστηρίου για να υπάρξει ανακοίνωση, επικοινωνία με το κοινό, η διάδοση ενός προστατευόμενου έργου θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τεχνικό τρόπο που να διαφέρει από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν ή να αφορά ένα διαφορετικό κοινό. Ένα κοινό που δεν έχουν λάβει υπόψη οι κάτοχοι του δικαιώματος δημιουργού στο παρελθόν όταν ενέκριναν την αρχική κοινοποίησή του. Σημείο 3. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε νομοθετικά αυτό που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όρισε σε ό,τι αφορά το linking and embedding. Η αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να αποκλείσει τα δύο αυτά μέσα να αποτελέσουν τρόπο επικοινωνίας με το κοινό, η κοινοποίηση στο κοινό και να μην συνδυαστούν με τη γενική υποχρέωση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 ε, αυτής της οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τον embedding, ο Ευρωπαίος δικαστής αναφερόμενος στα όσα ήδη αναφέρθηκαν στον τομέα του linking είπε ότι ότι δεν γίνεται ε, διαφορετική αναφορά από την αρχική, ούτε μεταφέρεται το έργο σε ένα διαφορετικό ε, κοινό. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτό, το δικαστήριο δήλωσε ότι η ένταξη στο, σε μία ιστοσελίδα ενό προστατευόμενου έργου μέσω της τεχνικής του embedding δεν μπορεί να θεωρηθεί ανακοίνωση, κοινοποίηση στο κοινό, γιατί το έργο δεν ε, ε, αφορά ένα νέο κοινό, ούτε κοινοποιείται με ένα διαφορετικό... Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Όλοι διάβασαν την γνωμοδότηση. Το θέμα είναι να υπογραμμίσεις ορισμένα σημεία. Γιατί καταλαβαίνεις αυτό είναι κάτι που δεν ήθιστε εδώ. Απλά και μόνο θα πρέπει να υπογραμμίσεις ορισμένα σημεία. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν ε, την δυνατότητα να διαβάσουν την γνωμοδότηση. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Από τη συνάντηση με τους χειώδεις συζητητές διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές πτυχές που δεν είχαν γίνει κατανοητές, γιατί μεταξύ των άλλων η γνωμοδότηση επειδή είναι σύντομη, δυστυχώς ε, παρακαλώ, θερμή παράκληση, σεβαστείτε το χρόνο σας. Σημείο 4. Η ίδια η έννοια της αναπαραγωγής θα πρέπει να επικαιροποιηθεί από τη στιγμή κατά την οποία οι δυνατότητες που προέρχονται σε επίπεδο ψηφιακό που σήμερα έχουν διάφορους τρόπους διανομής θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και την έννοια της αναπαραγωγής και να αποφευτούν οι επικαλύψεις. Συνεπώς, τυποποιώντας το δικαίωμα κοινοποίησης στο κοινό. Η έννοια αναπαραγωγής εντάχθηκε σε ένα αναλογικό πλαίσιο και στην ουσία δημιουργεί την επικάλυψη ενός έργου που ήδη έχει τη έγκριση. Σημείο 5. Εμείς δεν προτείνουμε τη δημιουργία νέων περιορισμών και εξαιρέσεων, αλλά την εφαρμογή τους στην υποχρεωτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλες οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί και ιδιαίτερα αυτέ που αφορούν την επιστημονική έρευνα, το σύστημα των ψηφιακών πληροθηκών θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη. Γιατί, γιατί ο, ο, ο χαρακτήρας της επαναχρησιμοποίησης είχε διπτές αρνητικές επιπτώσεις. Δεν υπήρχε νέος χαρακτήρας, δηλαδή δεν δημιουργήθηκαν διακρατικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργήθηκαν διακρίσεις. Όπως μου ζήτησε η πρόεδρος, θα ήθελα να καταλήξω κάπου. Όλα αυτά που αναφέρω τα πήραμε και από, την, από το, την πύλη ε, που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για να μπορέσουμε να ε, ασχοληθούμε με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ η Επιτροπή είπε σαφώ ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε αυτές τις αναφορές γιατί δημιουργούν διακρίσεις. Σημείο 6. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μία αντεμήνυμης εξαίρεση η οποία αφορά την, ε, το συνυπολογισμό νέων φαινομένων που προέκυψαν από, την ψηφία και από τις ψηφιακές ε, αλλαγές που έχουν γίνει. Κυκλοβάνει υπόψη τη χάρτα των θεμελιωδιών δικαιωμάτων σχετικά με την ερμηνεία ε, της μη διάκρισης. Αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει πάντοτε για να αξιολογείται στο φως συγκεκριμένων κριτηρίων που προβλέπεται από την οδηγία στο σημείο 55. Και αυτή η αναθεώρηση στηρίχθηκε από το την πύλη των Ηνωμένων Εθνών για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Εκεί λένε ότι ένα κλειστό κατάλογο δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο. Σημείο 7. ίσες απολαβές. απολαβές ε, αυτό είναι κάτι που γεννήθηκε σε αναλογικό πλαίσιο και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το σχέδιο μετα... Ε, αναθεώρηση της και τα όσα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση Διπιτορίνου του Ιανουαρίου του 2013 χρησιμεύει και στην εξασφάλιση μέγιστης διαφάνειας έτσι ώστε πολίτες και καταναλωτές να μπορέσουν να ε, ε, γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν. Μόνο έτσι θα μπορούσε κανείς να αποφύγει καιροσκοπικές συμπεριφορές. Θα πρέπει βεβαίως να εναρμονίσει τα κριτήρια να υπόψη το νέο ψηφιακό πλαίσιο. Σημείο 8. Τέλος. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις αρχές που αφορούν την ευθύνη των μεσαζόντων στο φως της κοινωτικής νομολογίας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι προβλεπόμενα από το σημείο 8 δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση με τα ε, θελμελιώδη δικαιώματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, ότι δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν από μια διοικητική αρχή και ότι θα πρέπει κατά αποκλειστικότητα να αποφασίζει το δικαστικό σώμα και κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι επικουρικές σε σχέση με την ε, καταστολή που προβλέπεται σε κάποια χώρα για να μην υπάρξει διακριτική ε, ε, μεταχείριση σε ό,τι αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε μια άλλη χώρα μέρος. Πέραν αυτού θα πρέπει να αφορούν τους πελάτες των παρόχων και όχι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτους όπως συμβαίνει τώρα. Θα ήθελα να τελειώσω. Ευχαριστώ ζητώντας την προ... Ε, για την προσοχή ελπίζω να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών και όχι των πολυεθνικών. Και δική μου ευχή είναι αυτή. Ελπίζω να εξισορροπηθούν τα διάφορα δικαιώματα, τα ε, δικαιώματα των δημιουργών και τα πνευματικά δικαιώματα να αναγνωριστεί η αξία τους γιατί και αυτό αποτελεί μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλοι μας θα καταβάλουμε μία προσπάθεια για να ε, πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Επιτρέψτε μου να δώσω σε δύο ακόμα συναδέλφους ε, το λόγο. Ο χρόνος μας πιέζει. Κώστερ και Ζουλό. Και θα τελειώσουμε. Α, ο συνάδελφος Καρβαρέσκη και θα έλεγα να κλείσουμε εδώ, αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτή τη συζήτηση. Ο συνάδελφος Τρούπελ. Θερμή παράκληση. Συνάδελφος Ρέιμον για την ομάδα των Πρασίνων. Διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Συνάδελφος Ρέιμον και Τρούπερ. Και οι δυο, και οι θέλετε να πάρετε το λόγο. Ωραία, ωραία. Τελειώνουμε εδώ. Ja, vielen Dank, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε και για την εκθεσή σας με την οποία κατέστησαν σαφή περισσότερα θέματα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Και εγώ, ε, μάλλον εγώ είμαι και μέλος ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, και <clears throat> Γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι γνωστή και η θέση της Επιτροπής Πολιτισμού για το θέμα των δικαιωμάτων του δημιουργού. <clears throat> Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς ως ε, μέλη αυτής της ε, Επιτροπής ενδιαφερόμεθα κυρίως να υπάρχει μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στους ε, δημιουργούς, τους ενδιάμεσους και τους χρήστες έχοντας καταρχήν κατά νου τους δημιουργούς. Και όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού θα πρέπει να μην έχουμε μόνο υπόψη μας τα θέματα των Χριστών, αλλά να μεριμνούμε το ότι σε ένα ψηφιοποιημένο κόσμο και οι δημιουργοί που αποτελούν την πηγή, την καρδιά του πολιτισμού και αυτοί θα πρέπει να στηρίζονται με δίκαιες αμοιβέ. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι ένα θέμα που νομίζω κυρίως ως Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο. Βεβαίως όλα αυτά σημαίνουν ότι η μεταρρύθμιση του δικαίου περί του δημιουργού, η μεταρρύθμιση αυτή θα συμβάλλει ε, στο να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια ε, σε επίπεδο χρηστών ε, και χρήσης του διαδικτύου και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γι' αυτό λοιπόν για μένα αυτό που παίζει ρόλο είναι να καταλήξουμε σε μια συμμαχία ανάμεσα στους δημιουργούς και τους χρήστες αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση ε, κατά την μεταρρύθμιση του δικαίου περί δικαιωμάτων δημιουργού αυτό θεωρούμε εμεί ότι είναι μια σημαντική πρόκληση Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε, συνάδελφος Ζηλό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κι εγώ. Έχω τρεις παρατηρήσεις που δεν αφορά την ε, παρουσίαση της συναδέλφου, αλλά τη γνωμοδότηση. Όσον αφορά το κείμενο αυτό καθεαυτό, εκπλήσωμαι και ανησυχώ γιατί λείπει από το κείμενο και αυτό είναι παράξενο. Λείπει από το κείμενο το θέμα των δημιουργών, ενώ είναι η πρώτη του οποίους αφορά αυτό το κείμενο, αυτή η γνωμοδότηση. Δεύτερον, υπάρχει ένας νομικός μηχανισμός που αναφέρεται στη γνωμοδότηση αυτή, που ουσιαστικά μοιάζει πολύ με τον αμερικανικό μηχανισμό του Fair Use, και που πραγματικά δημιουργεί προβλήματα στην νομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που κινδυνεύει να δυσκολέψει και τους δημιουργούς και τους καταναλωτές. Αυτός ο μηχανισμός fair ουσιαστικά προϋποθέτει ότι δεν γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων αν η χρήση είναι καλή ή όχι και ότι αυτό το θέμα μπορεί να επιληθεί μόνο ενώπιον των δικαστηρίων. Τρίτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι πέρα από την αναθεώρηση που προβλέπει η οδηγία του 2001, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να είναι ελεύθερα όσον αφορά τις επιλογές τους στην πολιτιστική τους πολιτική. Να ακολουθούν δηλαδή τις επιλογές τους και την παράδοσή τους και ανάγκες οι οποίες εκφράζονται και βεβαίως να τηρούνται οι εγκεκριμένες ε, διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε και να προσπιστούμε την πολυμορφία της δημιουργίας στην Ευρώπη. Θα υποβάλω λοιπόν μία τροπολογία έτσι ώστε να είναι πιο ισορροπημένη και πιο ορθή αυτή η γνωμοδότηση, αυτό το κείμενο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Και εγώ θα ήθελα εδώ να εκφράσω κάποιες ε, κριτικές ε, παρατηρήσεις όσον αφορά το ρόλο των δημιουργών, των καλλιτεχνών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά την στήριξη της ε, δημιουργίας και την χρήση. Υπάρχει η εμπορική και η μη εμπορική χρήση ενός έργου, μιας δημιουργίας. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη, για παιδαγωγική ε, χρήση. Τα, οι σύνδεσμοι για εμπορικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους μη εμπορικούς στο, ε, συνδέσμους, δηλαδή συνδέσμους για μη εμπορικό σκοπό. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το μπερδεύουμε. Ο δημιουργικός καλλιτεχνικός τομέας ε, στην ε, Πολωνία έχει αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και εδώ θα ήθελα να πω ότι η αρχή της εδαφικότητας παραδείγματος χάρη όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα και βέβαια κάποιος μπορεί να ξαναδεί αυτές τις αρχές, να τις επανεξετάσει, αλλά όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό. Έχει δίκιο εδώ η συγγήτρια, αλλά από την άλλη πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας όλα αυτά τα σημεία τα οποία σας προανέφερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριος Ρέιμεν και μετά η κυρία Τρούπελ και έτσι ε, θα κλείσουμε την παρέμβαση. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι σύντομο να σας πω ότι την έκθεση σε γενικές γραμμές την βρίσκω ιδιαίτερα ισόρροπη. Ε, Λείπουν εντάξει κάποια πράγματα, αλλά μπορεί κανείς να καταθέσει τροπολογίες. Στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, δεν είμαστε αρμόδιοι μόνο ε, για τα δικαιώματα των δημιουργών, αλλά και για τα δικαιώματα ε, των χρηστών όλων των πολιτών που καταναλώνουν πολιτισμό και που και αυτοί έχουν δικαιώματα. Στο μέλλον λοιπόν θα είναι συγκεχημένα τα όρια ανάμεσα σε δημιουργούς, μεσάζοντες ή ενδιάμεσους και Το νέο δίκαιο περί δικαιωμάτων δημιουργού θα πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνει υπόψη, δηλαδή να ενισχυθούν ε, τα δικαιώματα και των χρηστών και των δημιουργών. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα. Ε, παρότι μερικοί από την ε, βιομηχανία αυτή της κουλτούρας δεν συμφωνούν. Ε, κυρία Τρούπελ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όταν μιλάμε για εναρμόνιση των δικαιωμάτων του δημιουργού με άλλα δικαιώματα, ξεκινάμε από πολύ ψηλά. Ξεκινάμε από εξαιρέσεις και περιορισμούς. Καλά το κάνουμε αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να υπάρχει σωστή αποζημίωση για όλους τους δημιουργούς Όσον αφορά τα μουσεία, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, ε, τα πράγματα ξεφεύγουν και εκτός από γενικές εξαιρέσεις ε, θα πρέπει και εκεί να υπάρχει δυνατότητα της ε, ψηφιακής, της online πρόσβασης. Σημασία να δώσουμε μεγαλύτερη στην θέση των δημιουργών σε σχέση ή απέναντι, στον, απέναντι στους ενδιάμεσους. Η Κομισιόν δεν θέλει να πει τίποτα, γι' αυτό εγώ θα πω ότι αναμφίβολα θα υπάρξουν πολύ ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος είναι να υπάρχουν η σύμβαση που δίνουμε στην ε, καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Και θα ήθελα να παραμείνουμε στο σωστό τομέα όσον αφορά τις ε, προκλήσεις και τα δικαιώματα. Υπάρχουν λοιπόν τρία πράγματα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι και η ενδιάμεση. Και επ' αυτού ε, μην ξεχνάμε την πρωτοβουλία ο, με την οποία έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και ε, εδώ πλέον ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους γίγαντες του ίντερνετ που δεν είναι απαραίτητα Ευρωπαίοι και αυτοί ε, πραγματικά προδίδουν τα δικαιώματα του δημιουργού. Και το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια στη συζήτησή μας. Εν πάση αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ απλά θα ήθελα να συστήσω σε όλους να ε, προσπαθήσουν να βρουν αυτή την δύσκολη ισορροπία αλλά ξεκινώντας κυρίως από τις δικές μας τις αρμοδιότητες. Εμείς καλούμεθα να συντάξουμε μία γνωμοδότηση που να εντάσσεται στις δικές μας τις αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και βεβαίως και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και περνάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσια διάταξης που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει σχέση, ε, είναι το 9, έχει σχέση με τις ε, με το TTIP. Η συνάδελφος Τρούπελ είναι η συγγήτρια αυτής της τόσο σημαντικής γνωμοδότησης που ε, αφορά τη σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Γνωρίζετε ότι στόχος των πολιτικών ομάδων είναι να γνωμοδοτήσουμε επ' αυτού παρότι γνωρίζουμε ότι, και αυτό το είπαν και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και η Επιτροπή ότι όσον αφορά το TTIP, τη συμφωνία αυτή, εξαιρείται το ραδιοτηλεπτικό πεδίο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει αυτή την ε, έκθεση του Κοινοβουλίου, αυτή την τόσο σημαντική τοποθέτησή του, θα πρέπει να την πλαισιώσουμε και με τη δική μας τη γνωμοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι 9 Μαρτίου είναι η διορία ε, για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 16 Απριλίου ε, τα συνεδριάσουμε και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στη συνάδελφο κυρία Τρούιπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να πω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να προτείνει σαφείς ε, διατυπώσεις εδώ στην επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή ΙΝΤΑ όσον αφορά τα θέματα των ε, υπηρεσιών στον τομέα της ε, του πολιτισμού που μας αφορά. Και θα ήθελα εδώ να μιλήσω για την πολυμορφία, γιατί είναι σαφές ότι υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται σε αυτό τον τομέα. Αυτή η σύμβαση δείχνει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να ενισχυθούν και ότι πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητή η ιδιαίτερη ταυτότητα που θα πρέπει να περιέχεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στη γνωμοδότησή μας να φαίνεται με σαφήνεια ότι θέλουμε με δεσμευτικό τρόπο μία αναφορά στη σύμβαση της UNESCO και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την σύμβαση της UNESCO αλλά και τις συμφωνίες GAP καθότι εδώ θα πρέπει να στηρίξουμε τη ρύθμιση αυτών των ε, υπηρεσιών στο μέλλον με την λεγόμενη τεχνολογική ουδετερότητα που απαιτείται εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, να υπάρξει δηλαδή εδώ κανονισμός, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν οι υπηρεσίες αυτές, οι ψηφιακές, ε, σαν ψηφιακές υπηρεσίες και βλέπουμε εδώ ποια είναι η στάση των Αμερικανών, ομιλούν για ψηφιακά προϊόντα, εμπορικά δηλαδή προϊόντα. Εμείς θέλουμε αυτό να διαχωριστεί και θέλουμε σε κάθε περίπτωση να υπάρξει άλλη πολιτική και άλλη ρύθμιση για τα προϊόντα αυτά, για τις υπηρεσίες αυτές οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που εδώ δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει το θέμα της τιμής, της προκαθορισμένης τιμής του βιβλίου, κάτι που κατά την άποψή μας θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια στα πλαίσια της συμφωνίας TTIP. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όλα τα μέτρα στήριξης των ε, υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφέρονται ρητά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ε, δημόσια χρηματοδότηση και φυσικά σε κάθε περίπτωση το θέμα του ανταγωνισμού με την ιδιωτική εκπαίδευση και βεβαίως ότι αυτά είναι θέματα ακόμα ε, εθνικής αρμοδιότητας. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αυτά που εμείς προσφέρουμε εδώ για απελευθέρωση της αγοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε, μία, σε έναν κατάλογο αρνητικό, αυτά δηλαδή που δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην απελευθέρωση αγοράς. Και βεβαίως εδώ υπάρχει και όλη η εξέλιξη της τεχνολογίας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να μην είναι δηλαδή αποκλειστικός ο κατάλογος σε καμία περίπτωση. Και βεβαίως να δούμε τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό είναι η άποψη της πολιτικής μου ομάδας, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και γι' αυτό και δεν χρειάζεται σήμερα να τα αναφέρουμε. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η άποψη της πολιτικής μου ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική αυτή η γνωμοδότηση, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και προς το παρόν το υποστηρίζουμε. Ο συνάδελφος Μόργανο. Πολύ σύντομος. Σε ό,τι με αφορά θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Τρούπελ για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ανεξάρτητα από την πολιτική αξιολόγηση των ομάδων μας και ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση, Πιστεύω ότι θα δοθούν ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δεδομένο όμως ότι ο πολιτισμός δεν είναι πτυχές που δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εδώ. Νομίζω ότι κάνετε πολύ καλά που αναφέρεστε στη σύμβαση της UNESCO του 2005, γιατί στην ιστορία των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επιδοτήσεις στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού αποκλείονται από τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτή όμως η αντιμετώπιση δεν επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς που συνδέονται με τον πολιτισμό. Αναφέρομαι στις, ε, στα αρχεία, στα μουσεία, ε, αλλά δεν μπορώ να επεκταθώ για λόγους χρόνου. Η συνάδελφος Τρούπελ έχει θέσει ένα συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο τον εξήγησε όσα. Έκανε μία αναφορά στη γενική ρήτρα που θα πρέπει να ενταχθεί στην συμφωνία σε ό,τι αφορά τον ΚΑΤ και τη σύμβαση, σύμβαση UNESCO. Αν κατάλαβα καλά τα όσα την ευγένεια να πει συνάδελφος τις προηγούμενες μέρες κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το Διευθυντή Γενική Γενικής Διεύθυνσης Trade. Είχα την εντύπωση ότι κατάλαβα λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες που αφορούν το σημείο αυτό από την νομική άποψη. Πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια εμβάθυνση του θέματος από πλευρά τη Επιτροπής. Η κεντρική έννοια θα πρέπει να τονιστεί, να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, εμπορίου και επενδύσεων, σε ό,τι αφορά τις οπτοκουστικέ υπηρεσίες και τις ψηφικές υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την άλλη ρήτρα, την επαναπρόταση μιας γενικής ρήτρα που αφορά την παροχή υπηρεσιών για τους λόγους που η ίδια η κυρία Τρούπελ ανέφερε. Σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο θέματα αν δηλαδή είναι σκόπιμο ή δεν είναι σκόπιμο να συνταχθεί ένας θετικός ή ένας αρνητικός κατάλογος. Προσωπικά θα έλεγα ότι δεν έχω μία θέση εκ των προτέρων. Δεν ξέρω, θα ήθελα απλά και μόνο να πω ότι αν γινόταν μόνον ένας θετικός κατάλογος, αν το είχαμε κάνει πριν από πέντε χρόνια, δεν θα είχαν ε, δεν θα είχε ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογή συμφωνία η τηλεόραση ή streaming. Θέτω στον εαυτό μου το ερώτημα αν κατά κάποιο τρόπο είναι σκόπιμο να κινηθούμε προς την α ή προς τη β κατεύθυνση και ενδεχομένως ε, η Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει περαιτέρω στοιχεία. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μια γενικότερη αξιολόγηση το τελευταίο θέμα είναι ευαίσθητο. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι ένα θέμα οριζόντιο που αφορά όλη τη συμφωνία. Συνεπώς έχω τη βεβαιότητα και σας επιβεβαιώνω ότι σε, με αφορά ότι η ενδεχόμενη ένταξη ενός τέτοιου μηχανισμού θα μπορούσε να γίνει δεκτή υπό τον όρο ότι θα είναι ένα μεταρρυθμισμένο και σαφές μέσο. Πιστεύω ότι αν καταστεί αναγκαίο ή αν θεωρηθεί σκόπιμο, αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο, το να μπορέσουμε δηλαδή να προωθήσουμε εγγυήσεις οι οποίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ θα μπορούσα να παραθέσω ένα κατάλογο. Συγγνώμη, δεν, ο χρόνος μας πιέζει. Επιβεβαιώνω σε ό,τι με αφορά ο σκιώδης εισηγητής της ομάδας σοσιαλιστών την ε, στήριξή μου στη βασική ιδέα που την εξέφρασε η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Όλοι θέλετε να πάρετε το λόγο. Το επιβεβαιώνετε. Ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ε, πίεση. Ακολουθεί η συνάντηση των συντονιστών για αυτό το λόγο. Ερωτήσεις παρακαλώ. Α, Κέστερ, με συγχωρείτε. Κέστερ, Μίκα Φεράγια, Αντινόσκη. Παρακαλώ. Όλοι θέλετε να πάρετε το λόγο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Στο ένα λεπτό επάνω θα σας διακόψω. Η κυρία Τρίπελ υπέβαλε μια εξαιρετική έκθεση με πολύ σημαντικά σημεία που εμπεριέχονται. Στηρίζουμε λοιπόν αυτήν την πρότασή της. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, το θέμα της συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Δεύτερον, το θέμα των δικαιωμάτων δημιουργών στην υπηρετική Ευρώπη σε σχέση με αυτά που ισχύουν στις Ηνωμένε Πολιτείες στα πλαίσια της συμφωνίας. Τρίτον, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μέσω του TTIP να μην ανοίξουμε την πόρτα σε κάποιες απαγορεύσεις και περιορισμούς όσον αφορά την στήριξη των φορέων του δημόσιου τομέα. Πολύ σύντομα μια γενική παρατηρήση. Εγώ θα χαιρόμουν αν αυτό που έγινε και σε άλλες επιτροπές να δίναμε το λόγο όταν δεν υπάρχει χρόνος αρκετός για ομιλία στους κοιόδης εισηγητές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν. Δεύτερον, ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Τρίπελ για την εξαιρετική αυτή πρόταση έκθεσης και πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε όλες τις εξαιρέσεις στον τομέα του πολιτισμού και σε καμία περίπτωση να μην ξεχάσουμε το θέμα των υπηρεσιών του οπτικοακουστικού τομέα. Μια μικρή, μικρή προσθήκη θα ήθελα να κάνω επίσης στον κατάλογο αυτό Αυτή η γενική απόρριψη όσον αφορά την ε, επίλυση των διαφορών. Υπάρχει ένα σύστημα με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα που ουσιαστικά διέπει όλες τις συμβάσεις ή τις περισσότερες συμβάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών. Με διαφάνεια λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε να συνεχίσει να ισχύει αυτό το σύστημα, αυτή η διαδικασία και ενδεχομένω να προτείνουμε ενίσχυσή του, βελτίωσή του. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και νομίζω ότι μιλώ εδώ εξ ονοματο της, πολιτικη μου ομάδα. Δεν μπορούμε ειδικά για θέματα πολιτιστικά να αλλάξουμε τη διαδικασία όσον αφορά την επίλυση των διαφορών. Νομίζω ότι για τον τομέα του πολιτισμού θα ήταν πολύ καλύτερο αν παραμέναμε με τον κατάλογο τον αρνητικό. Νομίζω ότι αυτό το είχαμε πει και στην ε, συνάντηση και στην νόηση που είχαμε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται νέος κατάλογος, νέα ταξινόμηση αλλά να δεχτούμε αυτά που μέχρι τώρα έχουν καθοριστεί σαν τομείς και ενδεχομένως να προτείνουμε εμείς αυτόν τον αρνητικό κατάλογο. Αυτό είναι, αν θέλετε, οι δύο μοναδικές ε, παρατηρήσεις, ε, οι διαφορές που ήθελα να εκφράσω, κατά τα άλλα στηρίζω την πρόταση. Ο κύριε Ράιος, συνάδελφος Ντινόλφη, ο κύριος και οι δύο σκιώδεις συζητητές. Ένα λεπτό όμως παρακαλώ. Εγώ. Δεν υπογραμμίσαμε τις θετικές επιτυχίες στον τομέα του πολιτισμού. Για μας η πρόσβαση την εποχή του κομμουνισμού στην αμερικάνικη κουλτούρα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ένα μήνυμα ελευθερίας. Ενδεχομένω λείπει έστω και μία θετική πρόταση. Από την άλλη, η Ευρωπαίοι δημιουργοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Αμερικάνικη αγορά. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τον αποκλεισμό του οπτικο-ακουστικού τομέα. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, αυτές οι υπηρεσίες που έχουν ε, πολλές πολιτιστικές πτυχές. το σύστημα ESDS, επειδή υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών, Εγώ δεν θα ήμουν καταρχάς κατά της ιδέας, γιατί θα μπορούσε αυτό να σημαίνει μια ευκαιρία για να μπει κάποια τάξη σε αυτό το σύστημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σύντομα. Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο που υπάρχει γιατί δημιουργείται σύγχυση σε επίπεδο λεκτικό. Πολιτιστική υπηρεσία, τα οπτικοακουστικά είναι πολιτιστική δημιουργία. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Τρούπερ, αλλά βεβαίως τα λόγια ε, είναι λόγια. Δεν ξέρουμε τι είναι γραμμένο στις συνθήκες. Δεν ξέρουμε αν δημιουργικότητα και ευρωπαϊκός πολιτισμός, ιδιαίτερα των πιο μικρών χωρών, διακυβεύεται. Συνάδελφος Πίκελς. Α, με συγχωρείτε, έδωσα πρώτο λόγο στους χιλιάδες συζητητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, και εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο εξή ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο στη σκιώδη συγκήτρια. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Ε, τη γνωμοδότηση τη βρίσκουμε πάρα πολύ καλή, ισόρροπη, είναι κατά του SDS, αλλά και προβάλλει αιτήματα να υπάρχει έτσι ένας μικρός κατάλογος, ευσύνοπτος, με εξαιρέσεις. Ένα θέμα θέλω να δείξω, ότι εμείς θα θέλαμε να προβληθεί περισσότερο το θέμα της ε, εξαίρεσης των οπτικοακουστικών μέτρων. Ακούμε ότι υπάρχει έτσι ο δανασδητός χαρακτήρας του πολιτισμού, σωστό αυτό, αλλά γνωρίζουμε ότι ειδικά στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες τα οπτικοακουστικά μέσα είναι πολιτιστικό αγαθό και ως εκ τούτου προφανώς και θα ε, εμπίπτουν ε, στη συμφωνία TTIP. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να καταθέσουμε τροπολογίες έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να παρέμβετε και να κλείσουμε. Μισό λεπτό. Η Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Εσείς θέλετε κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ σύντομα, αν γίνεται, πάρα πολύ σύντομα, γιατί ξέρω ότι είστε υποποίηση. Εγώ απλά θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Το ένα εξ αυτών είναι η αναφορά στη σύμβαση της UNESCO. Αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι το εξής. Βεβαίως για κάποιον που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση της UNESCO, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως να είναι εύκολο να αναφέρεται σε αυτή τη σύμβαση. Και βεβαίως πολύ εύκολα μπορεί κανείς να εξαιρεί και αρχές που αναφέρονται σε αυτή τη συμφωνία με την UNESCO, δηλαδή την πολιτιστική διαφοροποίηση. Εδώ υπάρχει και εντολή του Συμβουλίου προς την Επιτροπή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το θέμα των ενισχύσεων που καταβάλλονται στον πολιτιστικό τομέα. Νομίζω κατά το παρελθόν έχω εξηγήσει ότι το θέμα των επιδοτήσεων κατά κανόνα δεν περιλαμβάνεται στις εμπορικές σχέσεις ούτε των ΗΠΑ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις επενδύσεις και την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή, αν τα κράτη-μέλη θέλουν με διακριτική μεταχείριση να συνεχίσουν να στηρίζουν πολιτιστικές ε, δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη τους ε, παρόχους ε, εκμάθησης γλώσσας, όπως ας πούμε το θεσμό Hochschulen στη Γερμανία, μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Η συμφωνία TTIP δεν αλλάζει τίποτα και οι ενισχύσεις δεν καλύπτονται από το κεφάλαιο απελευθέρωσης ε, παροχής υπηρεσιών ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και το τρίτο που αναφέρθηκε είναι εκείνο που έχει σχέση ε, με υπηρεσίες που έχουν πολιτιστική διάσταση. Όπως ξέρετε έχουμε κάποιο πρόβλημα με ένα τόσο ευρύ ορισμό γιατί στη Συμφωνία GATS υπάρχουν ε, πάρα πολλές επιφυλάξεις και εξαιρέσεις για βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Όμως, από την άλλη, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί, αν θέλετε, όσον αφορά τη σύσταση θεατρικών ομάδων ή μουσικών ομάδων. Αυτές λοιπόν οι υποχρεώσεις θεατρικών θεάσεων, πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να καλύπτεται από τη συμφωνία. Κατά παρελθόν προστατέψαμε πολλούς τομείς, τον οπτικοακουστικό πλήρως και κάποιους άλλους, ε, ε, όπου όμως τα κράτη-μέλη ε, έχουν αναλάβει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με βάση τη συμφωνία GATS. Η κυρία Τρούπελ Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για τις απόψεις τους και ε, θα τα βρούμε με τις τροπολογίες. Πολύ ωραία, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες. Ξέρω ότι η ημερησία διάταξή μας ήταν πάρα πολύ επιβαρημένη, αλλά τελικά μπορέσαμε να ακούσουμε κάποιες απόψεις για τα κείμενα άλλων επιτροπών που είχαν ε, φέρει πιο κοντά τις ε, καταληκτικές ε, προθεσμίες. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε. Θα ήθελα να σας παρακαλώσω να βγείτε ησύχως. Έχουμε τώρα τη συνεδρίαση των συντονιστών ίσως οι διερμηνείς μπορούν να μείνουν στην αίθουσα για να μας βοηθήσουν. Everything is very uncomplicated, so you just...